Ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ θερμά να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε χθες το βράδυ και να αφομοιώσετε και να χωνέψετε όλες τις εμπειρίες που βιώσαμε χθες. Ε, και σήμερα θα έχουμε ζωντανή αναμετάδοση από το διαδίκτυο και μάλιστα μπορείτε και με βίντεο κατά παραγγελία να ακούσετε τις διαλέξεις. Εκτός εθούσης, έχουμε φυλάδια με τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνίας και μάλιστα τα φυλάδια αυτά είναι μεταφρασμένα και στα τουρκικά και ρωσικά. Αν θέλετε μπορείτε να τα πάρετε. Χθε το βράδυ βρήκαμε και μία μηχανή κάνων ε, και που διπνήσαμε στην τραπεζαρία. Ιζαμπέλα, πήρε τη μηχανή. Όποιος την έχασε παρακαλώ να αποταθεί στην Ιζαμπέλα. Ο τελικός κατάλογος, ο οριστικός κατάλογος ε, με τους συμμετέχοντες ε, στο φόρουμ βρίσκεται πια και στην ιστοσελίδα μας, όποιος ενδιαφέρεται. Χθες ακούσαμε ότι η διερμηνία μπορεί να διδαχθεί, δεν είναι κάτι έφυτο, χρειάζεται πολύ στοχευμένη εξάσκηση Σήμερα όμως θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της διερμηνίας στον εγκέφαλο του διερμηνέα. Γιατί κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι οι διερμηνείς ε, δεν νοσούν από Αλσχάιμερ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πολύ το θέμα. Και μια και τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε τι τρέχει στο μυαλό του διερμηνέα. Ε, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ο επόμενος ε, καλεσμένος μας μπορεί πραγματικά να διερευνήσει τον εγκέφαλο του διερμηνέα. Είναι καλός φίλος ο επόμενος ομιλητής ε, της Γενικής Διεύθυνσης λέμε ο άνθρωπος εγκέφαλο και δεν τον ενοχλεί. Μάλιστα έκανε το διδακτορικό του στο Κέμπριτζ και ασχολήθηκε με τις επιστήμες του εγκεφάλου και είναι ερευνητής για τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Και το βασικό ερευνητικό του πεδίο αφορά τις ε, νευρονικές διαδικασίες και τη ε, διαδικασία της διερμηνίας καθώς και τις, επι... και τις συνέπειες της διαδικασίας αυτής στον εγκέφαλο. Παρακαλώ, ας χειροκροτήσουμε τον καθηγητή Άντελμαν Ερβέ Άντελμαν. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω την δυνατότητα να μοιραστώ την έρευνά μου μαζί σας θα σας παρουσιάσω αυτά τα οποία κάνουμε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης στα πλαίσια της Σχολής Μετάφρασης και Διαρμηνίας μαζί με το τμήμα της ιατρικής. Αυτό αφορά τις διαδικασίες της νευροβιολογικές στην ε, αυτόματη διαρμηνία, κάτι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Θα σας πω πώς χρησιμοποιούμε εμείς τον εγκέφαλο των διαρμηνέων είναι κάτι το πάρα πολύ... Είναι μια ικανότητα η διαρμηνία η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της μαθητείας και της πρακτικής. Είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο για μας έτσι ώστε να εξετάσουμε τις νευρονικές ζώνες όχι μόνο του γλωσσικού και γνωσιακού ελέγχου, αλλά μας επιτρέπει την δυνατότητα να ελέγξουμε και τις αλλαγές που γίνονται ε, στον εγκέφαλο του διερμηνέα, δηλαδή την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Μια και που θα σας μιλήσω για τον εγκέφαλο, να μου επιτρέψετε να σας προσανατολίσω επολίγων στα θέματα του εγκεφάλου. Βλέπετε εδώ στις οθόνες μία προβολή μέσα από το κρανίο του εγκεφάλου. Τον βλέπετε με πολλά χρώματα. Καταρχάς το μπλε είναι ο ηνιακός λοβός. Βλέπετε ότι αυτό καλύπτει την όραση, τα μηνύματα δηλαδή, τα οπτικά εκφράζονται και επεξεργάζονται από εκεί. Μετά η ζώνη που είναι σε κίτρινο είναι ο βρεγματικός λοβός που είναι πολύ σημαντικός για την αίσθηση ε, και την αισθητική δραστηριότητα αυτά τα οποία νιώθουμε στο σώμα μας σαν παράδειγμα και ασχολείται επίσης και καλύπτει τα θέματα της εστίασης προσοχής και της ε, διαλογικής συζήτησης μερικές φορές. Στα πράσινα βλέπετε τον κροταφικό λοβό, είναι σημαντικό για μας γιατί έχει σχέση με την ακρόαση. Ε, όλοι οι ήχοι ε, περνούν από τα αυτιά μας όπως επίσης και τα συναισθήματα και η μακροπρόθεσμη μνήμη και μπροστά έχουμε το μετοπιαίο λοβό ο οποίος είναι ο πιο σε εισαγωγικά σύγχρονος θα έλεγα στα πλαίσια της ερευνητικής μας διαδικασίας βλέπουμε εδώ τις λεγόμενες εκτελεστικές λειτουργίες. Τι είναι οι εκτελεστικές, είναι οι προχωρημένες γνωσιακές λειτουργίες, οι επιλογές, οι απαγορεύσεις, οι προγραμματισμοί ανάλογα με το δυναμικό περιβάλλον το οποίο είναι γύρω μας. Αυτό ελέγχει την κίνηση σαν παράδειγμα. Ε, στα πλαίσια των δύο αυτών λοβών, δηλαδή ε, του ε, Μετοπιέου και του κροταφικού, θα δούμε το ότι έχει σχέση με τη διερμηνία. Σας μίλησα για τις λεγόμενες εκτελεστικές διαδικασίες και λειτουργίες. Ε, μπορεί να είναι η εξής αν τις παρουσιάσουμε αναλυτικά. Υπάρχει το λεγόμενο switching το οποίο κάνει ο ε, διερμηνέας, η αλλαγή της γλώσσας δηλαδή. Υπάρχει ο έλεγχος σε σχέση με την προσοχή του, δηλαδή ο, ο διερμηνέας μοιράζει την προσοχή του ανάμεσα σε αυτό το οποίο ακούει και σε αυτό το οποίο λέει ε, υπάρχει το θέμα της ε, προσοχής για την αποφυγή των λαθών στην περίπτωση που προσπαθεί να αποφύγει ε, την, το λάθος. Υπάρχει και η, η διαχείριση της σύγκρουσης. Μερικές φορές ο διερμηνέας είναι πολύγλωσσος και χαρακτηριστικά όταν ελέγχουμε πάρα πολλές γλώσσες κάθε φορά χρησιμοποιούμε μία από τις γλώσσες αυτές. Όταν επικοινωνούμε με κάποιον προσπαθούμε να ομιλούμε τη σωστή γλώσσα. Υπάρχει μία διαδικασία σταθμιστική η οποία μας οδηγεί στη χρήση μίας γλώσσας, την επιλογή μίας γλώσσας. Ο διερμηνέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί όμως και δύο γλώσσες ε, πάρα πολύ συχνά και να αποφύγει αυτό το οποίο ακούει στην γλώσσα πηγής, κάτι το οποίο είναι δύσκολο μερικές φορές. Υπάρχει ακόμα και αυτό που ονομάζουμε η μνήμη της εργασίας. Εδώ αποθηκεύεται η πληροφορία. Ο διερμηνέας ε, σορεύει και αποθηκεύει την πληροφορία για να βγάλει το νόημα. Αυτή τη στιγμή βγάλει το νόημα, το μετατρέπει ε, προς την γλώσσα στόχο. Όλες αυτές οι διαδικασίες, οι εκτελεστικές λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσες, δεν αφορούν μόνο τη διερμηνία βέβαια, είναι σφαιρικές λειτουργίες και βλέπουμε ότι εδώ ε, οι δίγλωσοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μονόγλωσσους. Κάποιος ο οποίος ελέγχει πολλές γλώσσες σε καθημερινή βάση έχει κάποια πλεονεκτήματα στους τομείς αυτούς. Η μνήμη εργασίας στον Διερμηνέα βελτιούται. Αυτό δεν εκπλήσει κανένα γιατί ο Διερμηνέας είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με τη μνήμη του. Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι οι έμπειροι διερμηνείς στην ταυτόχρονη διερμηνία έχουν μια ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών η οποία είναι πλεονεκτική σε σχέση με αυτούς οι οποίοι απλά διδάσκουν ξένες γλώσσες ή είναι απλοί φοιτητέ ξένων γλωσσών έστω και πολύγλωση, όχι μόνο για να διατηρήσει στη μνήμη του μία σειρά αριθμών ή μία σειρά λέξεων, αλλά ακόμα και κάποιες γνωσιακές διαδικασίες που εξελίσσονται παράλληλα. Όχι μόνο αποθηκεύει δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα με την αποθήκευση επεξεργάζεται και την πληροφορία. Και όχι μόνο αυτό, ε, και αυτό εκπλήσει ακόμα περισσότερο, έχει και τη δυνατότητα να διαγράφει ε, τα στοιχεία τα οποία τον αποτρέπουν από το να συγκεντρώσει την προσοχή του. Έχουν μια αυξημένη αντίσταση στις εξωτερικές ενοχλήσεις θα έλεγα. Θα σας πω εδώ ε, ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο ε, θα σας δείξει πώς αποφεύγουμε τις εξωτερικές ενοχλήσεις. Βλέπετε το κέντρο της οθόνης με ένα σταυρό. Ξαφνικά βγαίνει κάτι που μας απασχολεί αριστερά και υπάρχει ένα κίνητρο από τη δεξιά πλευρά το οποίο όμως φάνηκε για μία μόνο στιγμή, για ένα δευτερόλεπτο. Αν εμείς έχουμε χάσει την προσοχή μας ε, λόγω της αριστερής εμφάνισης χάνουμε τη δεξιά, την στιγμιαία. Λοιπόν και αυτό έχουν, δείχνει ότι έχουμε αποτύχει. Οι διερμηνείς λοιπόν είναι πολύ καλύτεροι στο να αντισταθούν σε τέτοιου ε, είδους ενοχλήσεις αυτό βέβαια είναι στο οπτικό πεδίο, δεν είναι το πεδίο στο οποίο εργάζονται οι διερμηνείς. Οι διερμηνείς οξύνουν κάποιες ικανότητες που δεν αφορούν μόνο τη διερμηνία. Υπάρχουν και κάποια άλλα πλεονεκτήματα γνωσιακά των διερμηνέων που δεν περιμένει κανείς. Βλέπετε εδώ ε, κάτι το οποίο ονομάζουμε γνωσιακή ευελιξία ή γνωσιακή ελαστικότητα. Ε, πρόκειται για την επιλογή κάποιων καρτών. Υπάρχουν 128 στοιχεία, κάθε χαρτί, κάθε κάρτα μπορεί να γίνει αντικείμενο επιλογής είτε με βάση το χρώμα, είτε με βάση τον αριθμό των, ε, των σχημάτων, είτε με βάση τα ίδια τα σχήματα. Βλέπετε το ένα κόκκινο, το 2 με τον αριθμό 2 λόγω των αστέρων, 3 ε, και 4 κτλ. Βλέπετε ότι η αποστολή αυτή φαίνεται αρκετά απλή. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια κάρτες ε, με φυσιολογικό τρόπο μέσω του ενός ε, τεστ απλού να τοποθετήσουμε στη σειρά ανάλογα με την επιλογή ε, του κριτηρίου. Τι εννοώ με αυτό, θα πρέπει εμείς καθημερινά να ενημερώνουμε το σύστημα απεικόνησης το οποίο επεξεργαζόμαστε και οι διερμηνείς αυτό μπορεί να το κάνουν ταχύτερα από αυτούς που δεν έχουν εμπειρία στη διερμηνία. Η δυνατότητα που έχουν δηλαδή ε, να ενημερώνουν τις γνώσεις τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η άσκηση λοιπόν της διερμηνίας προκαλεί κάποιες γνωσιακές αλλαγές, θα πρέπει δηλαδή ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται. εμάς μας ενδιαφέρει αυτές τις γνωσιακές ε, πλεονεκτικές καταστάσεις να δούμε ε, σε ποιο βαθμό έχουν σημασία και στις διαδικασίες μάθησης της διερμηνίας. Έχει γίνει μια μελέτη η οποία γίνεται με μαγνητική απεικόνηση η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε στο εσωτερικό του εγκεφάλου την δραστηριότητα του εγκεφάλου ε, σε ένα φυσικά άνθρωπο εν ζωή και να εξετάσουμε ταυτόχρονα και τις αλλαγές στη μορφολογία του εγκεφάλου. Θα πρέπει να σας προσανατολίσω σιγά σιγά. Αριστερά βλέπετε δύο αναπαραστάσεις του εγκεφάλου. Από πάνω βλέπετε το αριστερό ημισφαίριο και κάτω το δεξί ημισφαίριο. Ε, το πράσινο μπλε χρώμα είναι οι δραστηριότητες του εγκεφάλου όταν ζητάμε κάποιες δραστηριότητες, όταν του ζητάμε να κάνουν το λεγόμενο shadowing, δηλαδή την, ταυτόχρονη επανάληψη. Απλά του ζητάμε να επαναλάβουν, όχι να κάνουν διερμηνία. Θα σας δείξω κάποιες άλλες ε, εικόνες, ανακόβουμε φέτες τον εγκέφαλο. Η δραστηριότητα αυτή της ταυτόχρονης επανάληψης αφορά την άρθρωση, την ακρόαση, την συγκέντρωση και όλες τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εξελίσσονται στα πλαίσια της ταυτόχρονης επανάληψης. Εδώ με, την πορτοκαλί, ε, με τους πορτοκαλί κύκλους βλέπετε τον χώρο του Μπροκά που είναι πολύ σημαντικός για τον έλεγχο της άρθρωσης και την παραγωγή της ομιλίας. Ο δεύτερος πορτοκαλής ε, κύκλος είναι ο χώρος του Βερνικέ και αυτός έχει σχέση με την ομιλία είναι κάτι που έχει όμως σχέση και με την κατανόηση, δηλαδή η κατανόηση που μετατρέπεται σε ομιλία. Και στις δύο τελευταίες πορτοκαλία απεικονίσεις βλέπετε το λεγόμενο κινησιακό συμπληρωματικό χώρο, κάτι το οποίο έχει σχέση με τα συναισθήματα. Δεν είναι μόνο θέμα εκτέλεσης συγκεκριμένων προγραμμάτων κίνησης, αλλά είναι και θέμα προγραμματισμού και ανείχνευσης λαθών όταν κάνουμε μια κίνηση και δεν πετυχαίνουμε να την κάνουμε όπως θέλουμε, ε, οι περιοχές αυτές ευαισθητοποιούνται πλήρως. Τι συμβαίνει τώρα στον εγκέφαλο όταν ε, προσθέτουμε την πολυγλωσσική ε, δραστηριότητα μέσω της διερμηνίας. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει. Στο κόκκινο εδώ αριστερά βλέπετε ακριβώς το τι ενεργοποιείται για την αποστολή της διερμηνίας, για τη δραστηριότητα της διερμηνίας ότι είναι σε μπλε και ε, πράσινο είναι σημαντικό για την επανάληψη και είναι φυσικά ε, απαραίτητο και για τη διερμηνία. Υπάρχει όμως και μια επιπλέον γνωσιακή αποστολή, ένα επιπλέον γνωσιακό βάρος το οποίο έχει άμεση σχέση με τον γλωσσικό έλεγχο. Βλέπετε λοιπόν ένα δίκτυο εδώ το οποίο ανήκει στο σύστημα το οποίο ασχολείται με τον προγραμματισμό ε, και ταυτόχρονα έχουμε και ένα τμήμα του χώρου Μπρόκα που ασχολείται με την σημασιολογική κωδικοποίηση. Ξεκινώντας από το κέντρο του εγκεφάλου βλέπουμε στο πάνω αριστερά μέρος το πράσινο μπλε που έχει μεγάλη σημασία με την έννοια ότι κάνει τις επιλογές όταν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες σαν παράδειγμα σε μια άλλη μαγνητική τομή Βλέπετε ότι το κόκκινο εδώ είναι πολύ μικρότερο. Έχουμε τον λεγόμενο κωδικοποιημένο πυρήνα. Είναι το λεγόμενο, θα έλεγα, chez nous, les humains, mais aussi chez les lézards, chez les rongeurs, qui ne sont évidemment pas linguistiques. nous permet de choisir des mouvements, d'effectuer des mouvements και αν πρέπει να αλλάξουμε την κίνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να περάσουμε πάντα από τον ερπετιαίο αυτό πυρήνα. μια μικρή ε, δομή, ένα μικρό όργανο το οποίο ελέγχει την κίνηση περισσότερο. Βλέπετε ότι μιλάω πάρα πολύ για κίνηση και όχι τόσο για γλώσσα. Ε, οι όροι μερικές φορές είναι γλωσσικοί, μερικές φορές δεν είναι. Εδώ ελέγχεται η κίνηση ουσιαστικά ε, και ακριβώς αυτή η κίνηση είναι το σημαντικό. Εδώ βλέπετε τον πυρήνα κοντέ που είναι ο κερκοφόρος πυρήνας. Ε, πρόκειται για μια, ε, μια λειτουργία η οποία ελέγχει και αυτή εν μέρη την κίνηση, ασχολείται όμως και με τα θέματα της μάθησης, των κινήτρων, ε, της επιλογής και της επιλογής των σχημάτων και των προτύπων μερικές φορές των επαναλαμβωμένων. Το θέμα είναι πώς ο εγκέφαλος ελέγχει το ταυτόχρονο της διερμηνίας, πώς ακούμε και μιλάμε. Υπάρχει ένα τμήμα του εγκεφάλου το οποίο το ελέγχει αυτό. Το έχουμε ελέγξει και έχουμε δει ότι σε αυτήν εδώ την μαγνητική τομή ότι υπάρχουν δύο ζώνες πολύ σημαντικές ακριβώς δίπλα από τον κερκοφόρο είναι ε, το κωδικοποιημένο αυτό κέλυφος το οποίο επιτρέπει ε, την τέλεση περίπλοκων ε, ε, δράσεων που έχουν όμως γενικό χαρακτήρα. Σαν παράδειγμα γνωρίζετε πολλές φορές από την οικογένειά σας την ασθένεια του Πάρκινσον. Τα συμπτώματα αυτά προέρχονται από βλάβες σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου. Έχουμε να κάνουμε με κάτι που δεν έχει σχέση με την διαρμηνία, αλλά έχει σχέση περισσότερο με τον έλεγχο της κινητικότητας και τον έλεγχο τον γνωσιακό. Έχουμε ελέγξει επίσης και το θέμα της εκπαίδευσης και της πρακτικής. Έχουμε την τύχη να δουλεύουμε με ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ Βλέπουμε το πρότυπο λειτουργίας στην διερμηνία μετά την εκπαίδευση. Βλέπετε εδώ μια διαφορετικού προσανατολισμού τομή. Μια τομή η οποία δείχνει ακριβώς μετά την εκπαίδευση, μετά την πρακτική που έχει υπάρξει μια αλλαγή. Βλέπουμε πάντα ότι είναι ο κερκοφόρος πυρήνας αυτή η αλλαγή. Θα σας εξηγήσω ε, το τι γίνεται σε αυτόν τον πυρήνα η έκφραση των αλλαγών οι οποίες οφείλονται στην εκπαίδευση, στην πρακτική, οδηγούν σε μία μείωση των δραστηριοτήτων κάποιων τμήματων του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης πρακτικής. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η δομή αυτή η οποία δραστηριοποιείται και αυτή τη στιγμή καθίσταται αυτόματη η διερμηνία αυτή γιατί ε, κάποια άλλα τμήματα του εγκεφάλου έχουν διαφορετικού τύπου αντιδράσεις. Ε, το τμήμα αυτό αφού μαθαίνει να κάνει κάτι το κάνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο, δραστηριοποιείται πολύ λιγότερο και αυτό απελευθερώνει τις άλλες δυνατότητες που έχει ο διερμηνέας για να βελτιώσει την επίδοσή του. Η εμπειρογνωμοσύνη επίσης έχει σχέση με τον κερκοφόρο πυρήνα. Υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στα δικά μας αποτελέσματα και αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί σε άλλους τομείς όπως τους μουσικούς, αυτούς που παίζουν σκάκι, κάποιους αθλητές και κάποιους αθλητές του γκολφ ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς αυτός ο κερκοφόρος πυρήνας ενεργοποιείται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης βλέπουμε αν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές μορφολογικές, διαρθρωτικές, λόγω ακριβώς της διαδικασίας εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι η δραστηριότητα, η απεικόνηση της δραστηριότητας στα πλαίσια του, α, της αλλαγής του όγκου του εγκεφάλου όπου εμπλέκεται ο εγκέφαλος στην διερμηνία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά θα σας πω ότι υπάρχουν ε, ε, εμπλοκές πάλι τομέων όπως του κερκοφόρου πυρήνα που επηρεάζουν την εκμάθηση της διαδικασίας της διερμηνίας. Συνοπτικά εμείς λέμε ότι η διερμηνία εξερτάται από νευρονικά δίκτυα τα οποία εμπλέκονται στη γνωσιακή διαδικασία ελέγχου, ότι η άσκηση της διερμηνίας φαίνεται να αυξάνει την αποτελεσματικότητα αυτών των ιδίων συστημάτων. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε, έχουμε κάποιες προοπτικές στην έρευνα στον τομέα αυτό, θα συνεχίσουμε την έρευνα αυτή με πιο έμπειρους διερμηνείς, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα συγκεντρώνοντας μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία. Προσπαθούμε να δούμε τις επιπτώσεις της άσκησης της γερμηνίας στις γνωσιακές ικανότητες μέσω των αλλαγών στον εγκέφαλο στις οποίες αναφέρθηκα ήδη και σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα για την διασύνδεση διερμηνίας και άλλων δραστηριοτήτων θα δούμε τι γίνεται με την ομοιότητα κάποιων εγκεφαλικών προσαρμογών που προκαλούνται από τη διερμηνία. Και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι η λεγόμενη διαρθρωτική συνδεσιμότητα, δηλαδή όλες οι συνάψεις, όλες οι επικοινωνίες οι οποίες γίνονται στον εγκέφαλο και οι οποίες εκφράζουν τη διασυνδεσιμότητα. Βλέπετε αυτά τα μακαρόνια, αυτό το σπαγγέτι είναι νευρώνες οι οποίοι συνδέουν μεταξύ τους τα τμήματα του εγκεφάλου. Αυτό είναι θεμελιώδες για τη λειτουργία του εγκεφάλου γιατί η καλωδίωση αυτή ακριβώς είναι αυτή που καθορίζει τις ικανότητες επεξεργασίας και τις ικανότητες της, της, της διάθεσης για ε, επεξεργασία. Είμαστε ικανοί με την μέθοδο αυτή να κάνουμε μία τομή in vivo του εγκεφάλου σε συγκεκριμένα τμήματα για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τις συνάψεις. Βλέπουμε εδώ δύο ε, σύνολα, δύο δεσμίδες βλέπουμε το φεσό αρκιουέ, δηλαδή την τοξοειδή δεσμίδα η οποία συνδέει το τμήμα που έχει σχέση με την παραγωγή της ομιλίας και το τμήμα που έχει σχέση με την κατανόηση της ομιλίας. Φαίνεται ότι αυτή η δεσμίδα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με την λεγόμενη μνήμη εργασίας, γιατί εκεί βγαίνει και παράγεται η ηχό που συνδέει την αντίληψη της ομιλίας με την παραγωγή της ομιλίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκτυο το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε μια σωστή αναπαράσταση της δραστηριότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ επίσης και το Εθνικό Ελβετικό Ταμείο Έρευνας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ. Thanks Σας ευχαριστούμε θερμά, Dr. Αντελμαν. Και παραμείνετε παρακαλώ στο Προεδρείο, γιατί μετά την παρουσίαση την επόμενη, που θα γίνει από δύο καλεσμένες, θα έχουμε γύρω ερωτήσεων και απαντήσεων. Ε, φαντάζομαι θα διαπιστώσει κάποιες ομοιότητες μεταξύ μουσικών και διερμηνέων ε, σε ό,τι αφορά τις ε, διεργασίες και τις αλλαγές στον εγκέφαλο. Και θα κάνουμε μία άσκηση πριν ο Φίλιπ βρίσκεται ήδη εδώ και θα ενεργοποιήσει το σύστημα της ψηφοφορίας, οπότε ε, επειδή είναι μυστική ψηφοφορία θα πρέπει να βάλετε το χέρι στη μηχανή και να πατήσετε το συν για το ναι και το μείον για το όχι. Ποιος είναι υπέρ ε, ενός δωρεάν γεύματος μετά την συνεδρίαση. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας, να δούμε τα αποτελέσματα παρακαλώ Φίλιπ. Δεν προλάβατε να ψηφίσετε. Θα ήθελα να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Δεν πρέπει να πιέζετε τις ταμπέλες αλλά και τα εικονίδια, αλλά τα κουμπιά που βρίσκονται μέσα και θα τα πιέσετε προς εσάς. Μπορούμε τώρα να δούμε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Λειτουργήσε το σύστημα, ψήφισαν σχεδόν όλοι. 142. Η πραγματική ερώτηση όμως που θέλω να κάνω τώρα είναι ποιοι από εσά τραγουδάτε ή παίζετε ένα μουσικό όργανο. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίε. Πόσοι από εσά ε, είτε παίζετε όργανο είτε τραγουδάτε. Άρχεται η ψηφοφορία το πράσινο κουμπί για το ναι και το κόκκινο για το όχι. Μπορούν και οι συνάδελφοι από τις καμπίνες με τα χέρια, να σηκώσουν τα χέρια όσοι τραγουδάνε, παίζουν κάποιο όργανο. Ψηφίσατε όλοι. «88 έχουν κάποια σχέση με τη μουσική. Πολύ καλό σκορ. Μήπω έχουμε και κανένα διευθυντή ορχήστρα εδώ, έστω και ερασιτέχνη. But musical conductors, yes. No, but we have at least a good score. Ε, τουλάχιστον έχουμε αρκετούς μουσικούς, μπορεί να έχουμε διευθυντές, ορχήστρας πολλούς. Αλλά αυτή ήταν η εισαγωγή για τις επόμενες παρουσιάσεις. Καταρχήν η δόκτωρ Μαγδαλένα Ολιβέρα αποφύτησε ε, από το Πανεπιστήμιο σε, σε ε, διερμηνία και μετάφραση και μετά ε, ε, εργάστηκε στη Γενέβη και έκανε το διδακτορικό της με θέμα τη μουσική εκτέλεση και την, και την ε, ταυτόχρονη διερμηνία υπό τη σκοπιά όμως της πολυδιεργασίας. Και έχουμε και την Ναταλή που Ναταλή Λουαζό που είναι φρύλας διερμηνέας και κάνει το δακτορικό της τώρα στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Πριν έκανε μάστερ για τις μεσονικές σπουδές και επίσης πραγματοποιεί έρευνα σε θέματα πολυδιεργασίας για διευθυντές ορχήστρας και ταυτόχρονες ε, διερμηνείς. Διερμηνείς μάλλον σε ταυτόχρονη διερμηνία. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ για την καταπληκτική αυτή η παρουσίαση, δεν μπορούσα να περιμένω τίποτα καλύτερο ασφαλώς. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λοιπόν σήμερα οι δυο μα, για να περιορίσουμε και την πολυεπιτέλεση που θα κληθείτε εσεί να κάνετε, θα είναι να εξηγήσουμε πώ λειτουργεί η πολυεπιτέλεση, η multitasking. Θα μπορούσα πρώτα να σα δείξω μία ταινία και μετά ε, να σα βάλω να ακούσετε μια ραδιοφωνική εκπομπή, θα ήταν πιο εύκολο ίσω. δεν θα είχαν καμία σχέση μεταξύ του, αλλά ο άλλο τρόπο να σα δείξω πώ λειτουργεί αυτό είναι να βάλετε τα ακουστικά σα. Γιατί εκεί έχουμε του 30 έξι διερμηνείς, 33 διερμηνείς οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, το multitasking, πολύ επιτέλεση. Έχω και έναν ε, διαγωνισμό για τους διερμηνείς προς όλους, άλλωστε, να μου βρείτε το ισοδύναμο του multitasking στα γαλλικά. Εγώ λέω execution de tâche επιτέλεση πολλαπλών ε, καθηκόντων, αλλά ε, ελήψη μίας και ενίας λέξεως, ξαναπέφτω στο, στη μία λέξη, την αγγλική, το multitasking. Αν λοιπόν θέλετε να συναντήσετε το Θεό λένε, καθίστε σε μια ήσυχη και μιλήστε του. Εάν θέλετε να τον δείτε όμως, στείλτε ένα SMS την ώρα που οδηγείτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δουλεύει σε κάθε περίπτωση, αλλά εν περιπτώσει μπορεί κανείς να δοκιμάσει. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι δεν φαίνεται να είμαστε εκ των προτέρων προγραμματισμένοι ως όντα για την ε, πολυδιεργασία. Τι κάνουμε λοιπόν όταν κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και για να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μπορώ να συγκρίνω μουσικούς και διερμηνείς, αυτό θα το κάνει μετά η Μανταλένα και μετά θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα εάν μπορεί κανείς να γίνει καλός στην πόλη διεργασία ή στη διερμηνία ή τη μουσική. Αντίστοιχα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε διάφορους τύπους διεργασία, διάφορου τύπου προσέγγισης, διάφορου τρόπου προσέγγισης. Έχουμε παραδείγματι αυτό που αναφέρουμε συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωση ω media multitasking, πολυδιεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωση. Ε, Φερρυπίν κάποιο που δουλεύει στον υπολογιστή του, στέλνοντα ταυτόχρονα μηνύματα στου φίλου του, παρακολουθώντα το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η πολυδιεργασία σε ε, μέσα μαζική ενημέρωση. Επίση, οι γραμματεί στα ε, γραφεία πολύ συχνά χωρίς να είναι αυτό το καθήκον τους, ε, η περιγραφή του έργου τους, αναγκαστικά κάνουν πολλή διεργασία γιατί την ώρα που, γράφουν, που δακτυλογραφούν μια επιστολή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορεί να πρέπει να πατήσουν στην πόρτα κτλ. Και βεβαίως έχουμε και τη διερμηνία η οποία καλύπτει όλα αυτά τα, όλες αυτές τις λειτουργίες που σας περιέγραψα νωρίτερα και επίσης τους εναέριους ελεγκτές αν ξέρατε τι καλούνται να επιτελέσουν οι αέριοι ελεγκτέ, ίσω να διστάζατε να παίρνετε το αεροπλάνο, αλλά σα διαβεβαιώ ότι το καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Και η διερμηνία λοιπόν και η πολυδιεργασία είναι κάτι το σχετικά εύκολο να εξασφαλιστεί. Κάποια καθήκοντα δηλαδή μεταξύ του ε, σχετικά λίγο πολύ και έτσι διευκολύνεται η δυνατότητα να επιτελέσουμε περισσότερε ε, εργασίε ταυτόχρονα. Αλλά βέβαια είναι ασφαλέ το συμπέρασμα ότι κάνουμε λιγότερο καλά και λιγότερο γρήγορα όταν προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Προφανώ, αν μου ζητήσετε εμένα την ίδια παρουσίαση που σα κάνω τώρα, να σα την κάνω ταυτόχρονα πρέπει να στείλω και ένα SMS από το τηλέφωνό μου, μάλλον θα αρχίσω να μιλάω πιο αργά, ή μπορεί να χάσω λίγο τον ερμό μου, ή μπορεί να στείλω το SMS μου γεμάτο σφάλματα. Άρα η, μολ, η, η <laughs> πόλη διεργασία είναι ένα πολύ περίπλοκο έργο και σημαίνει πολλά, ε, πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα και παράλληλα. Εδώ λοιπόν, όταν κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έχουμε αυτή την ιδέα που είδαμε και νωρίτερα και που έχουμε διαπιστώσει και σε σχέση με τα μηχανήματα εχθές, με την παρουσίαση, παράξενο αυτό, είναι η γνωσιακή επιβάρυνση. Ο γνωσιακός φόρτος, ο οποίος έχει ένα ένα βαθμό αυτοματοποίησης επειδή ελέγχεται από τις πρωτόγονες ε, πτυχές του εγκεφάλου μας επιτρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα ορισμένα πράγματα. Να μιλούμε παραδείγματι. Από την άλλη υπάρχουν άλλα, άλλες εργασίες, άλλες διεργασίες, οι οποίες συνεπάγονται κάτι διαφορετικό. Όταν ακούει κανείς τη μητρική του γλώσσα ή αν ακούει μια ξένη γλώσσα, καταρχάς δεν χρειάζεται την ίδια προσπάθεια, το έργο αυτό. Από την άλλη όμως αν πρέπει να το συνδυάσει και με ένα, μια άλλη προσπάθεια, οι αυτοματισμοί δεν είναι οι ίδιοι. Αν προσπαθήσετε να κάνετε μια συνομιλία την ώρα που μιλάτε ή που έχετε την προσοχή σας στραμμένη σε κάτι, αλλά ακούτε ξαφνικά κάποιος να μιλάει τη μητρική σας γλώσσα, κάτι θα καταγράψετε αυτομάτως. Αν πρόκειται για ξένη γλώσσα θα πρέπει να είναι πολύ πιο συνειδητή η προσπάθεια για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και εδώ προφανώς θα δούμε και τις συνέπειες ως προς την διερμηνία. Θα μου πείτε ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να, με, μεταφράζει κανείς από την γλώσσα α, από την κύρια μετρική γλώσσα, προς τη γλώσσα β. Ε, προαιώνια η συζήτηση, αλλά ναι, ας πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σωστά η μετάφραση από την α στη β, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τη δυσκολία της απόδοσης σε μια γλώσσα β και τον περιορισμό του λεξιλογίου όπου βεβαίω θα συμφωνήσουμε όλοι πω η δίγλωση μπορεί να έχουν πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα δεδομένο ο συνδυασμό και αυτοματοποιημένο. Για όλα λοιπόν τα καθήκοντα, για όλε τι εργασίε που δεν είναι αυτόματες ή αυτοματοποιήσιμε, έχουμε κάποιου μηχανισμού οι οποίοι όμω πάντα έχουν του περιορισμού και τα προβλήματά του. Έχουμε την, εργασία, την ε, μνήμη εργασία μα επιτρέπει δηλαδή να κρατάμε στο μυαλό μα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ενό έργου. Αυτό σημαίνει, έχει όμω περιορισμού, δηλαδή δεν μπορώ να περάσω εύκολα από το ένα έργο στο άλλο. Φανταστείτε μια γραμματέα η οποία πολύ γρήγορα θα, θα φτάσει στο σημείο κορισμού και θα είναι και μονομανής μαζί. Αυτό θα σήμαινε να έχουμε μια περιόριστη επιβάρυνση της μνήμης εργασίας. Ταυτόχρονα όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθεί κανείς την πληροφορία, οπτική, ακουστική, ακόμη και συνδυασμό με το προσωπικό με, με, τα προσωπικά στοιχεία του, του εγκεφάλου, τη διαχείριση του στρες, παραδείγματι, να υπάρχει αυτός ο φόρτος, να εντοπιστεί, να αναγνωριστεί, να αποφασίσουμε αν θα τον διαχειριστούμε, να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα τον διαχειριστούμε, να αποφασίσουμε με ποια σειρά θα αντιδράσουμε, να μετατρέψουμε αυτό σε μια άλλη πληροφορία και να περάσουμε στο switching, που επίσης στα γαλλικά μπορούμε και shifting, δηλαδή με τη μεταφορά στην άλλη γλώσσα. Και αυτό σημαίνει ότι και ταυτόχρονα έχουμε μια προσοχή περιορισμένη προς κάθε κατεύθυνση. Ε, ας δούμε λίγο τους ε, ταχυδακτυλουργούς. Τα κόλπα, τα ταχυδακτυλουργικά, στηρίζονται ακριβώς στην αδυναμία του ανθρώπου να αντιληφθεί κάθε τι. Δηλαδή ε, εστιάζουμε την προσοχή μας σε κάτι και χάνουμε ένα στοιχείο από κάπου αλλού. Και επίσης δεν μπορούμε να περνάμε την προσοχή μας από τη μία στην άλλη πολύ γρήγορα. Φερρυπίν, ένας ανώτατος, ένα ανώτατος τέλεχος το οποίο χωρίς να αναθέτει σε κανέναν κατώτερό του καθήκοντα, τα αναλαμβάνει όλα αυτά, μάλλον η γραμματέας του αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα του ίδιου του στελέχους και, τον, ε, και τα εκτελεί. Εδώ η επεξεργασία μπορεί να καλύπτει περισσότερα καθήκοντα, αλλά μόνο επιφανειακά, όπως όταν παίζουμε στο παιχνίδι ηλεκτρονικά η συγκέντρωση όμως μπορεί να αναφέρεται μόνο σε ένα αντικείμενο. Όταν κάνουμε λοιπόν την πολυδιεργασία, περνάμε πολύ γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο με την προσοχή μας συνειδητά στραμμένη προς ένα πράγμα. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ασχοληθούμε οπωσδήποτε και απόλυτα με δύο πράγματα. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, περνούμε από το ένα, πηδάμε από το ένα στο άλλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Ε, κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ πιο εύκολο όταν έχουμε αυτοματοποιημένα καθήκοντα. Οι παρατηρήσεις που έχουμε από τον εγκέφαλο δεν μας καθησυχάζουν ιδιαίτερα. Καταρχάς έχουμε ε, μία σύραγγα, ένα σημείο κυκλοφορικής, ε, κυκλοφοριακής συμφόρησης στο προμετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, όπως είδαμε και νωρίτερα σχέση με τις γνωσιακά καθήκοντα και έχουμε έναν κεντρικό μηχανισμό ο οποίος κατεργάζεται εξεργάζεται όλες τις πληροφορίες, απολύτως όλες τις πληροφορίες ε, που, λαμβάνουμε, που λαμβάνει. Άρα καλό είναι αυτό γιατί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους σπόρους ανάλογα με το τι χρειάζεται το κάθε καθήκον, αλλά από την άλλη για να μπουν στο ε, σημείο αυτό του εγκεφάλου όλες οι πληροφορίες πρέπει να πάρουν σειρά η μία μετά την άλλη. Και προφανώς από τη στιγμή ε, ε, μεταξύ της στιγμής που θα γίνει η επιλογή και θα δοθεί εντολή για την αντίδραση, βρισκόμαστε σε ένα σημείο συμφόρησης, στενοπό. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνο, λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος του βραχικυκλώματος. Και όμως βλέπουμε το παράδεξο ότι εδώ ε, αντί για κίνδυνο βραχικυκλώματος, ή μάλλον στην περίπτωση του βραχικυκλώματος γίνεται πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μπορεί να περάσει πληροφορία από κάπου αλλού και όχι από αυτή τη σύραγγα. Βρίσκει ένα καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί την πληροφορία. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ο διαχωρισμό. Εάν κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα, εστιαζόμενοι σε δύο διαφορετικού στόχου ταυτόχρονα, εάν δηλαδή έχουμε ένα στόχο και μόνο θα επικεντρωθεί ολόκληρος ο εγκέφαλος σε αυτό το στόχο. Εάν έχουμε δύο στόχους, ο εγκέφαλος θα αρχίσει να χωρίζεται, το κάθε, μυστέριο θα ασχολείται με έναν στόχο, πολύ πρακτικό αυτό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα είναι λιγότερο αποτελεσματική η αξιοποίηση των πόρων μας, για να μην πω ότι θα γίνει αν βάλουμε και τρίτο στόχο μπροστά μας, γιατί εδώ έχουμε μελέτες οι οποίες μας δείχνουν γεωμετρική επιτρία, δηλαδή άνοδο του ποσοστού σφάλματος ε, και γενικά των εμπλοκών μεταξύ των τριών κομματιών που διαχειρίζονται την πληροφορία και το έργο. βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να διαχειριστούμε ένα σύνολο καθηκόντων ως μια, ένα ενιαίο καθήκον για όσους διδάσκουν τη διερμηνία είναι πιο εύκολο να εξηγήσετε στον φοιτητή ότι είναι πολύ σημαντικό και να καταλάβεις και μετά να μεταφράσεις και να τα πεις πολύ σωστά. Αν τα πείτε όμως έτσι χωριστά, μπορείτε να τους οδηγήσετε σε αμηχανία και φόβο. Εάν τους πείτε, κοίταξε να εξηγήσει το, το μήνυμα, να περάσει το μήνυμα σωστά, τότε καταλαβαίνουν πολύ καλύτερο, εν, καλύτερα εν γέννη οι φοιτητέ και μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την εντολή κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ για να δείξουμε πόσο περιορισμένες είναι οι δυνατότητες μας και οι μηχανισμοί μας. Δεν ισχύει πάντα αυτό γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια άτομα που φαίνεται να έχουν δυνατότητα πολυδιεργασίας κατά πολύ υπέρτερη του μέσου όρου χωρίς να έχουν ιδιαίτερο ιστορικό με βάση ένα κοινό δείγμα ε, πληθυσμού έχουμε ένα 2% με πολύ καλύτερες δυνατότητες σε πολυδιαργασία, ακόμη δε περισσότερο Βέβαια πρέπει να είναι κανείς ε, στην, στο βασικό του καθήκον καλός ξεκινώντας, να το συνδυάσει με κάποιο άλλο, με κάποια άλλη εργασία. Ε, αλλά έχουν λιγότερη δραστηριότητα στην, στον, στην περίφημη αυτή σύραγγα, στο Σύμβολο Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και ταυτόχρονα μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τα, ε, τις παρενοχλήσεις. Ε, μπορούμε λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα τώρα, με όλα αυτά τα μειονεκτήματα να φτάσουμε, να βελτιώσουμε την πολυδιεργασία. Μπορούμε οποιοδήποτε καθήκον ή έργο να το συγκρίνουμε με κάποια άλλα και έτσι να αναπτύξουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε περισσότερα καθήκοντα ταυτόχρονα. Είναι κάτι στο οποίο έχουν οι διερμηνείς γνωσιακό πλεονέκτημα αλλά που μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε άλλες πολλαπλές ε, ε, διεργασίες ε, στη ζωή ή τι είδους παράγοντες ή μεταβλητές μπορεί να βοηθούν κάποιον να βελτιώσει την πολυδιεργασία του. Αυτά θα μας τα πει η Μαγδαλένα Ολιβέηρα με μια σύγκριση των ικανοτήτων πολυδιεργασίας με, ε, με, στους διερμηνείς από τη μία και στους μουσικούς από την άλλη. Merci beaucoup, Nathalie. Σε ευχαριστώ, Ναταλή. Θα περάσω τώρα στα αγγλικά και θα σας ανακοινώσω τα συμπεράσματα της έρευνας που έκανα στο διδακτορικό μου στην οποία προσπάθησα να βρω τις ομοιότητες μεταξύ μουσικής εκτέλεσης και διερμηνίας. Κυρίως ε, στη μουσική με συνοδεία και στην ταυτόχρονη διερμηνία. Γιατί λοιπόν διάλεξα αυτές τις δύο δραστηριότητες. Πρώτα απ' όλα σπούδασα στο 2 πιάνο. Ήμουν πιανίστας, ε, έπαιζα, έπαιξα πιάνο και συνόδευα άλλους μουσικούς, ε, σαξοφωνίστες, βιολιστές και είχα την αίσθηση ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο κεφάλι μου, στον εγκέφαλό μου. Δεν ξέρω, ίσως ήταν ο κερκοφόρος πυρήνας που μου έκανε τη ζημιά. Άρχισα λοιπόν ε, να προβληματίζομαι γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω κάποια έρευνα. Και η μουσική που παίζουν μουσική με συνοδεία πρέπει να ακούν τους υπόλοιπου μουσικούς που εκτελούν τα δικά τους μουσικά κομμάτια, να κάνουν μια επεξεργασία των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο αυτό που ακούν και ταυτόχρονα μετά να παράγουν τη δική τους μουσική εκτέλεση. Και οι διερμηνείς που κάνουν ταυτόχρονη διερμηνία πρέπει να ακούν τον ομιλητή στην γλώσσα πηγή, να επεξεργάζονται τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και κατόπιν να μεταφέρουν το μήνυμα στη γλώσσα στόχο. Για να συγκρίνουμε τώρα με συστηματικό τρόπο αυτές τις δύο δραστηριότητες θα σας παρουσιάσω τρία σενάρια σύγκρισης. Νομίζω ότι κάποιος χθες θέση 83 ρώτησε τι γίνεται με την πρόβα και τη σημασία της πρόβας. Όντως η μουσική κάνουν ε, επανειλημμένα πρόβες στα κομμάτια τους. Μεγάλη εξάσκηση. Εγώ θα επικεντρωθώ όχι σε μια μουσική που έχει μάθει κανένας ε, εκ των προτέρων, αλλά σε πρίμα βίστα ανάγνωση παρτιτούρας και σε αυτοσχεδιασμό μουσικό. Καταρχήν έχουμε εδώ ανάγνωση παρτιτούρας πρίμα βίστα από ε, πιανίστες και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τη σύγκριση μεταξύ πρίμα βίστα ανάγνωση παρτιτούρας και πρίμα βίστα διερμηνίας Βλέπετε το σκορ λοιπόν στην οθόνη και βλέπετε για πρώτη φορά στη ζωή σας αυτό, αυτή την οθόνη και θα πρέπει ταυτόχρονα να επεξεργαστείτε τα στοιχεία, δηλαδή είτε να παίξετε την παρτιτούρα είτε να μεταφράσετε αυτό που βλέπετε. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές γιατί στην ε, διερμηνία αβίστα θα πρέπει να γίνει και η μεταφορά του μηνύματος από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου. Αυτό δεν συμβαίνει τόσο στη μουσική. Εκτός αν αλλάζετε και τον τόνο όταν διαβάζετε την παρτιτούρα. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Το δεύτερο σενάριο σύγκρισης αφορά την ε, μουσική με συνοδεία και με ταυτόχρονα, ταυτόχρονη ανάγνωση παρτιτούρας για πρώτη φορά και την ε, ταυτόχρονη διερμηνία με κείμενο. Έχουμε λοιπόν ε, μία πληροφορία είτε ε, σε κείμενο είτε προφορική και όταν έχουν το κείμενο μπροστά τους οι διερμηνείς ταυτόχρονα το ελέγχουν και το ίδιο και οι μουσικοί όταν διαβάζουν μια παρτιτούρα. Δηλαδή συγκρίνουν αυτό που έχουν στην παρτιτούρα με αυτό που ακούν από τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Αν εγώ παίζω πιάνο και ε, έχω και κάποιο φλαουτίστα δίπλα μου, μπορεί να μην τηρήσει πιστά την παρτιτούρα. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να παρακολουθήσω τις αλλαγές και να προσαρμοστώ στις αλλαγές που κάνει στο μουσικό κομμάτι. Βλέπετε αριστερά στην οθόνη ε, υπάρχει ένα ε, πορτοκαλί τμήμα που δείχνει μια σημαντική διαφορά γιατί στη μουσική με συνοδεία ένα σημαντικός παράγοντας είναι ότι προσθέτετε το δικό σας ήχο τη δική σας μελωδία στον ήχο που παράγουν άλλα μουσικά όργανα ώστε να βγαίνει ένα αρμονικό μελωδικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν συμβαίνει στη διερμηνία. Δεν χρειάζεται να συντονίζετε τη, τη φωνή σας ως διερμηνέας με τη φωνή του ομιλητή. Οπότε στη μουσική, όταν κάποιος παίζει, κάποιοι μουσικοί παίζουν ταυτόχρονα, έχουμε μια συνολική ακέρη ε, προσοχή γιατί πρέπει να συντονίσουμε και να συμπεριλάβουμε σε ένα μελλοντικό κομμάτι όλους τους μουσικούς. Ενώ στους ε, διερμηνείς έχουμε κάποια παράγωγη προσοχή γιατί ουσιαστικά αποσπούμε την προσοχή μας από το αρχικό μήνυμα. Υπάρχει διαφορά λοιπόν μεταξύ μουσικών και διερμηνών στο σημείο αυτό. Το τρίτο σενάριο σύγκρισης είναι ο αυτοσχεδιασμός αυτοσχέδια μουσική με συνοδεία και αυτοσχέδια διερμηνία. Εδώ έχουμε μόνο το προφορικό input, την επεξεργασία και το τελικό προϊόν, το output. Βλέπετε εδώ το πιο σημαντικό, το κόκκινο τμήμα στην ε, αριστερή πλευρά, στο συγκεκριμένο σενάριο και ο φλαουτίστας και ο πιανίστας και ο σολίστ δηλαδή και αυτός που τον συνοδεύει παράγουν, δημιουργούν νέο υλικό. Ε, αυτό το κάνουν και οι διερμηνείς μερικές φορές. Παράγουν νέο υλικό. Αυτά είναι θεωρητικά σενάρια. Γιατί ήθελα να θέσω μία ερώτηση, να, προβληματισμό, να προβληματιστώ. Γιατί και η μουσική και οι διερμηνείς χρειάζεται να κάνω πολλή διεργασία, να κάνουν ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών εργασιών. Γι' αυτό και πήρα το τεστ αυτό που το σχεδίασε η Ναταλή Λουαζό και η Σόφη Χέγγελ, μια άλλη συνάδελφος. Και εκεί διαφορετικές ομάδες συμμετόχων έκαναν ταυτόχρονα διάφορα πράγματα. Έπρεπε να διαβάσουν φωναχτά ένα κείμενο και ταυτόχρονα άκουγαν δυνατά μπιπ ε, και πιο σιγανά μπιπ και έπρεπε ταυτόχρονα να μετρήσουν πόσα μπιπ δυνατά και πόσα μπιπ πιο σιγανά άκουγαν και ταυτόχρονα να δουν αν καταλάβαιναν και το μήνυμα του κειμένου που διάβαζαν. Όταν τελείωσαν την ανάγνωση του κειμένου δυνατά, έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το περιεχόμενο του κειμένου. Εδώ προσπάθησα να λάβω υπόψη κάποιες γλωσσικές μεταβλητές, για παράδειγμα το βαθμό γνώσης ε, το, της γλώσσας, την έκθεση στη γλώσσα, πόσα χρόνια είχαν μείνει στη χώρα και κάποιες μουσικές μεταβλητές που είναι αυτές που επεξεργάστηκα και προηγουμένως ε, στο μοντέλο μου, δηλαδή η πείρα τους διαβάζουν παρτιτούρες πρίμα βίστα, σε μουσική με συνοδεία, σε συμμετοχή σε ορχήστρα, χρόνια σπουδών μουσικών και το καθεξής. Και Έχουμε εδώ τα σκορ με τρεις διαφορετικές ομάδες. Γενικώ διαπιστώσαμε ότι η μουσική ήταν καλύτερη από τους διερμηνείς σε ορισμένα θέματα και οι διερμηνείς σε άλλα. Σε σχέση με, το, με την ομάδα ελέγχου. Βέβαια η ομάδα ελέγχου δεν ήταν ομοιόμορφη, ομοιογενής. Γιατί στην κόκκινη στήλη έχουμε κάποια κάποιους που είχαν και μουσικές γνώσεις. Ενώ τα μπλε είναι εκείνο που, που είχαν ελάχιστες γνώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ομάδα με τους διερμηνείς και για την ομάδα με τους μουσικούς. Οι κόκκινοι στήλη είναι όσοι είχαν πολύ καλές ε, γλωσσικές γνώσεις και είχαν και καλύτερες επιδόσεις από τους άλλους οι διαφορές ε, μεταξύ των τριών ομάδων από στατιστική άποψη είναι μελιτέες, που σημαίνει ότι η ομάδα, η έννοια της ομάδας δεν είναι σημαντική. Αυτό που βλέπετε όμως με τις κόκκινες στήλε είναι ότι η μουσική φαίνεται, οι μουσικές γνώσεις φαίνεται να έχουν κάποιο σχετισμό, κάποια αντιστοιχεία. Οπότε θεώρησα το όλο δείγμα ως αδιέρετο. Πήρα ολόκληρο το δείγμα των 53 συμμετεχόντων και εξέτασα τους σχετισμούς, τις αντιστοιχίες. Εκεί είδα κάποιες πολύ σημαντικές και αλληλένδετες μεταβλητές. Οι μουσικές μεταβλητές ε, σχετιζόταν με το σκορ των ε, όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι οι πιο σχετισμένες ε, μεταβλητές το τελικό σκορ ήταν η, το, η ανάγνωση αβίστα και η εκτέλεση σε μία ορχήστρα, η συμμετοχή σε μία ορχήστρα. Και βλέπετε από το μοντέλο ότι μπορούσαμε ακόμη και να προβλέψουμε το σκορ του υποψηφίου ανάλογα με τα χρόνια είτε ενασχόλησης ε, με τη μουσική, της εξάσκησης ή του διαβάσματος παρτιτούρας. Και βλέπετε ότι είχαμε μια νοδική πορεία των αποτελεσμάτων που ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, αυτό ήταν ένα πιλωτικό τεστ και στην περίπτωση αυτή διερωτήθηκα αν η μουσική ή όσοι έχουν μουσικές σπουδές ή κάποιο μουσικό υπόβαθρο είναι πιο ικανοί στην πολυδιεργασία από ό,τι άλλοι. Ή ήταν ικανη για διερμηνία. Τους έκανα μια σύντομη προφορική παρουσίαση χωρίς κείμενο και ε, όσοι λάβανα μέρος έπρεπε να, να κάνουν διερμηνία του κειμένου χωρίς να έχουν προηγούμενη πείρα σε διερμηνία. Παρουσίασα ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε και στην πρώτη άσκηση, στο πρώτο πείραμα. Τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέροντα, γιατί είδα κάποιους σχετισμούς μεταξύ της γλώσσας πηγής και το επίπεδο της γλωσσομάθειας της πρώτης ξένης γλώσσας, της γλώσσας από την οποία γινόταν η δερμηνία και το σκορ, το τελικό του σκορ. Οπότε όσοι είχαν τρίτο, ήταν στο τρίτο επίπεδο είχαν μέχρι πέντε, στο τέσσερα ήταν μέχρι δύο και στο πέντε μέχρι τριάμιση. Όταν ήταν κάτω από το επίπεδο 3 δεν ε, γίνονταν δεκτοί καν. Καταλήγω λοιπόν σε κάποια συμπεράσματα. Όσοι ε, είχαν κάποια μουσική παιδεία είχαν καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την πολυδιεργασία. Βέβαια δεν ήταν ε, μουσική αυτή η άσκηση αυτό το πείραμα και πολύ πιθανόν η μουσική αυτή ε, έπρεπε να μεταφέρουν αυτές τις, τις ικανότητές τους για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του πειράματος. Βέβαια το θέμα είναι ήταν επίκτητε αυτέ οι ικανότητε πολυδιεργασίας, Δηλαδή τι απόκτησαν κατά τη διάρκεια των μουσικών σπουδών, που άρα σημαίνει ότι μπορούν να διδαχθούν αυτέ οι ικανότητε πολυδιεργασίας, αυτέ οι δεξιότητε. Ή ήταν κάποια ταλέντα έμφυτα ή κάποιες δεξιότητες ε, multitasking είναι έμφυτες, αλλά στην έρευνά μου δεν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Εγώ απλώς ε, παρατήρησα ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ότι όσοι είχαν μεγαλύτερη γλωσσομάθεια είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Αν και επαναλαμβάνω, οι στατιστικές διαφορές ήταν αμελητές. Και επίσης οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις. Και εδώ όμως δεν είχαμε σημαντικές διαφορές στατιστικά. Σε ό,τι αφορά το πιλωτικό τεστ για την ε, ταυτόχρονη διερμηνία, ο μόνος σχετισμός που έκανα ήταν ότι όσοι έλαβαν μέρος με καλύτερη γλώσσα ε, της πρώτης ξένης γλώσσας είχαν καλύτερες επιδόσεις. Στην περίπτωση αυτή η μουσική δεν ήταν καλύτερη, οπότε αυτό μπορεί να οφείλεται είτε επειδή στο ότι κάποιες δεξιότητες είναι χαρακτηριστικές συγκεκριμένου κλάδου και άρα μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά στο συγκεκριμένο πείραμα δεν ε, ασχολήθηκα με φοιτητέ του οδείου αλλά απλώ με ανθρώπου που είχαν κάποιε μουσικέ σπουδέ και κάποιου όχι. Όχι όμω πολύ προχωρημένε. Σε άλλη έρευνα θα πάρω φοιτητέ του ΟΔΙΟ. Και επίση ε, είχαμε κάποιε άλλε τάσει. Τι θετικέ τάσει από του μουσικού και επίση τι καλύτερε επιδόσει των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες. Ε, ε, αλλά επαναλαμβάνω οι διαφορές αυτές ήταν αμελητές. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της δικής μου έρευνας. Ευχαριστώ. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπάρχει όταν βλέπει το θέμα κανείς του multitasking είναι να δει αν υπάρχει η δυνατότητα αυτών των ικανοτήτων. Αν μπορούμε σαν παράδειγμα να παίζουμε βιολό, βιολί διερμηνεύοντας ή να στέλνουμε SMS οδηγώντας. Ας κοιτάξουμε λίγο εδώ τα αποτελέσματα της εισαγωγικά εκπαίδευσης προπόνησης η ε, προπόνηση επιτρέπει να συνδυάσει κανείς διαφορετικές αρμοδιότητες. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς πολύ εύκολα να κάνει την ίδια στιγμή. Για το λεγόμενο media multitasking, ε, η συνεχής αλλά και όχι σε βάθος προσοχή και συγκέντρωση, μπορεί κανείς να συνδυάσει πολυτροπικά κίνητρα, αλλά όχι να κάνει σημαντικότερη και γενικότερη πρόοδο και να ασχοληθεί με δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Γιατί έχουμε δυσκολία εκεί να διαχειριστούμε ε, τα μηνύματα τα οποία μας κάνουν να αποκλίνει η προσοχή μας από αυτό το οποίο κάνουμε. Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι ασκούνται σε επίπεδο διαλογισμού, οι οποίοι μαθαίνουν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα πράγμα και όχι στα υπόλοιπα. Κάτι το οποίο θετικά τους βοηθάει στον τομέα της μαθητείας, της εκμάθησης καλύτερα. Τώρα για τη διαδικασία, το τι παρατηρούμε στον εγκέφαλο. Ο αυτοματισμός καθιστά την αποστολή σε σχέση με τις σκόπιμες δυνατότητες συλλογής πόρων και τον οποίων όμως η επεξεργασία γίνεται λιγότερο συνειδητή. Περνάμε από διαδικασίες του εγκεφάλου πολύ λιγότερο πρωτόγονες και αυτό καθιστά το multitasking πολύ πιο αποτελεσματικό εσείς σηκώνετε το τηλέφωνο, θέλετε να καλέσετε κάποιον, το κάνετε όμως με πολύ αυτόματο τρόπο και ξεχνάτε ταυτόχρονα ότι το κάνετε και κάνετε και άλλα πράγματα μαζί. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν και το βλέπουμε αυτό στη μουσική. Ό,τι είναι παραγωγός ήχου κίνηση είναι αυτοματοποιημένη μπορεί κάποιος να συμμετέχει παίζοντας ένα όργανο σε ένα κονσέρτο και να κάνει και πράξεις αριθμητικές. Αυτό μπορεί να το συνδυάσει. Δεν θα χρησιμοποιήσει λάθος νότες, δεν θα αλλάξει ρυθμό. Ενώ αντίθετα, και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι κάποια συνειδητά ερεθίσματα είναι πολύ σημαντικά, ότι, ε, ότι καθορίζει το εκφραστικό της προσπάθειας την οποία κάνει ε, καταπίπτει τη στιγμή που προσθήκεται ε, μια δεύτερη αποστολή. Το στρες σαν παράδειγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια επιπλέον ε, απασχόληση και δραστηριότητα. Τώρα, η σκόπιμη ακριβώς επεξεργασία της πληροφορίας είναι αλήθεια ότι γίνεται πιο γρήγορη. Έχουμε την δυνατότητα λόγω της άσκησης να επεξεργαζόμαστε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό έχει άμεση σχέση με την ενίσχυση της διαδικασίας επανάληψης της άσκησης. Τώρα, για το multitasking πάντα, ε, υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί κανείς να κινητοποιεί την προσοχή του σε διαφορετικά επίπεδα. Από τη μία συνειδητοποίηση των στίμουλη και ταυτόχρονα ταχύτητα επεξεργασίας κάνετε ένα υπολογισμό, μία πράξη ε, και έχετε κάποιους αριθμούς μπροστά σας. Αν αντικατασταθούν οι αριθμοί από χρώματα πάλι θα τα καταφέρετε εφόσον είστε Αυτό σημαίνει ότι ε, κάποιες ε, διαδικασίες οι οποίες γίνονται στα πλαίσια του multitasking μπορεί να τύχουν ενός προγράμματος εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. Δυνατοτήτων μάλλον. Λοιπόν τώρα αν μπορούμε να διδάξουμε το multitasking πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με τρόπο γενικά πρακτικό, μεταφέρσιμο. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις συνοδητές, συνειδητές ενέργειες από τη μία και τις αυτοματοποιημένες από την άλλη. Να διαχειριστούμε τις διαθέσιμες ορευμένες ικανότητες η προσοχή λειτουργεί με αυτοματισμούς πάρα πολύ συχνά και στους διερμηνείς. Καμιά φορά βέβαια πιστεύει ο διερμηνέας για πέντε λεπτά την ώρα που δουλεύει ότι το κάνει με αυτόματο τρόπο και σαν να ξυπνάει κατά κάποιο τρόπο από αυτό το οποίο κάνει κάποια στιγμή. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι παράλληλα με αυτό τον αυτοματισμό πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα κρίσης και λήψης απόφασης και πρέπει να αλλάξει κανείς ανάλογα με το πλαίσιο κτλ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών συνδυασμών στην διερμηνία. Οι δυσκολίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους ανάλογα με τον ομιλητή, ανάλογα με το πλαίσιο, την ακουστική κτλ. Δεν υπάρχει μία ενιαία δραστηριότητα δηλαδή. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι όταν κάποιος εργάζεται σε ένα πλαίσιο δεν είναι σε θέση να το μεταφέρει αυτόματα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Έχουμε ανάγκη δηλαδή από συγκεκριμένα πλαίσια. Λοιπόν, και μια άλλη, αν θέλετε, δυσκολία είναι να μπορεί κανείς να εκπαιδεύσει τους διερμηνείς ε, με προσαρμόσιμο τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με αποτελεσματικό τρόπο. Τελείωσα. Νομίζω ότι μετά από αυτά που είπα θα στέλνουμε σε μέσο ένα στον άλλο οδηγώντας, χωρίς όμως να συναντήσουμε και το Θεό παράλληλα. Ευχαριστώ πολύ Μάγδα, Ναταλή. Περάστε παρακαλώ στο Προεδρείο. Ίσως θα μπορούσαν ε, τα παρόντα εδώ πανεπιστήμια να, να παίρνουν για, τα... για τις σχολές διερμηνίας φοιτητές από τα μουσικά σχολεία. Πάντως με χαρά βλέπω αυτή την πολύ καλή έρευνα. Είναι και η νονά τους, η νονά των ερευνητριών. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Η Μπάρμπαρα Μόζερ Μέρσερ είναι ερευνητρία από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, είναι η ιδρύτρια του InZone. Μπάρμπαρα, ακούσαμε αυτά τρία παραδείγματα έρευνας. Χτες ακούσαμε ότι για να γίνει κανείς ε, άρτιος εκτελεστής θα πρέπει να κάνει πολλή εξάσκηση. Πώς τα συνδυάζουμε λοιπόν όλα αυτά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Προσκαλέσατε τη ομάδα. Με μεγάλη χαρά ήρθα να παρουσιάσω τη δική μας θεώρηση στην διαδικασία αυτή εκμάθησης της ερμηνείας και θα ήθελα να πάω λίγο πίσω και να μοιράσω τα σχόλιά μου τα εισαγωγικά σε δύο κομμάτια. Καταρχάς, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του να αντιληφθούμε πόσο περίπλοκο είναι το έργο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το ανέφερε και ο Αλέξης. Για μας, στη διερμηνία, το να αξιολογήσουμε δηλαδή ποια είναι τα έξω σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο εγκέφαλος ή να αντιληφθούμε τις προσαρμογές τις οποίες πρέπει να προβεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος ο εγκέφαλος του διερμηνέα και κυρίως μέσα σε ένα περιβάλλον ε, προηγμένης τεχνολογίας. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε, πόσο προσαρμόσιμο είναι ο εγκέφαλος και βέβαια μια βάση συγκρίσεως που θα πρέπει να εξασφαλιστεί, αυτό που είδαμε προς το τέλος, να καταλάβουμε καλύτερα άλλα έργα ή άλλες δεξιότητες και τις μεταβλητές που μπορούν να εντοπιστούν, να απομονωθούν και να ε, χρησιμεύσουν για τη σύγκριση μεταξύ των διαφορών εργασιών. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και σε αυτό οφείλει και την ύπαρξη του τομέα μας. Πρέπει να αντιληφθούμε δηλαδή τη βασική, τις βασικές δομές. Αλλά όπως και χθες ακούσαμε από τον Άντερς και είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του στη συνέχεια. Πρέπει να καταλάβουμε και την απόκτηση μιας δεξιότητα πώς λειτουργεί αυτή Πώς μπορούμε δηλαδή, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας ο τελικός, να μορφώσουμε, να εκπαιδεύσουμε μια, μια σειρά, μια γενιά διερμηνέων που εν τέλει θα κάτσουν στην καμπίνα και θα μπορέσουν να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε καλά αυτές τις δομές, γιατί μόνο αναλύοντας τη διαδικασία απόκτησης με πολύ μεγάλη προσοχή και όχι μόνο από, άποψη συμπεριφοράς, αλλά από γνωσιακή θεώρηση μπορούμε να αντιληφθούμε την απόκτηση άλλου τύπου δεξιοτήτων. Και εδώ είναι το κρίσιμο για μένα. Εκεί που έχει φτάσει δηλαδή η έρευνα στη διερμηνία. Γιατί, Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μια ενδοσκοπική προσέγγιση, κοιτούσαμε προς τα μέσα, πώς μπορεί η έρευνα να ενημερώσει την πρακτική, να βελτιώσει την πρακτική. Τώρα όμως θα πρέπει να ε, προασπιστούμε τη θέση και το ρόλο μας στο πανεπιστημιακό γίγνεσθε και πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο και σχετικά γρήγορα όπου το να γίνεται κατανοητή η λειτουργία της διερμηνίας ως περίπλοκου καθήκοντος θα έχει σημαντικό ενδιαφέρον και για, άλλα, για άλλους τομείς της επιστήμης. Όπου δηλαδή οι ερευνητές θα μαθαίνουν από μας γιατί η περιπλοκότητα των έργων που επιτελούμε δεν υφίσταται αλλού, δεν μπορεί να βρεθεί αλλού. Αρχίζουμε δηλαδή να προσφέρουμε επιστήμη, ε, απαντήσεις στην επιστήμη, αρχίζουμε να κοιτάζουμε συγκρίνοντας τις ανθρώπινες δεξιότητες, να αποκαλύπτουμε κάποιες από τις κοινέ μεταβλητές και ενδεχομένως σε κάθε τομέα βέβαια της επιστήμης ακούγεται η ενιαία ή η οικουμενική θεωρία και ίσως να φτάσουμε και εκεί τελικά μέσω της ερμηνείας. Αλλά πάντως αναζητούμε κοινέ παραμέτρους που επιτρέπουν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων και έτσι μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε τις διαφορετικές δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο. Αυτά εισαγωγικά για να συνδυάσω τα όσα ακούσαμε από τις σημερινέ τοποθετήσεις και παρουσιάσεις σήμερα και να σας επιτρέψω να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας. Έχει ουσιοδέστατη σημασία για την κατάρτιση, γιατί την τελική παιδαγωγική προσέγγιση με βάση μια επιστημονική γνώση και όχι μια καταπροσέγγιση ε, επιλογή του εμένα έτσι μου φαίνεται καλύτερο, μπορούμε να την προωθήσουμε έτσι μόνο και βεβαίως όπως είπα θα κερδίσουμε και θα πρόσπιστούμε έτσι τη θέση μας στον χώρο των πανεπιστημίων που επίσης με μεγάλο κόπο αναζητούμε. Ευχαριστώ πολύ. Περίπλοκη η ε, απάντησή μου, λέει η κυρία Μόζερ. Ευχαριστώ πολύ. Διεξοδική απάντησή σου. Μπορείτε να απευθύνετε τι ερωτήσει σα στου τρει ερευνητέ μα, είτε στην κυρία Μπάρμπαρα Μόζερ Μέρσερ. Παρακαλώ, φαντάζομαι ότι θα έχετε πολλέ ερωτήσει, να επικεντρώνεστε στην πιο ουσιαστική και συγκεκριμένη. Καλημέρα και ευχαριστώ για τις τρεις αυτές πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ιδιαίτερος με ενδιαφέρει η κατάρτιση των διερμηνέων στην ε, γλώσσα των κοφαλάλων. Ε, θέλω λοιπόν να μου πείτε εάν έχετε κάποια προσέγγιση ε, και μελέτη της οπτικής παραμέτρου σε αυτή την κατάρτιση και επίσης η οπτική προσέγγιση στον διερμηνέα η επαφή με το, κοινό, με το ακροατήριο, με τους εκπροσώπους σε τελευταία ανάλυση, γι' αυτό έχουν τζάμι οι καμπίνες. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι μία ε, εργασία διερμηνίας που περνάει μέσα από οθόνες επιβαρύνει με πολύ μεγαλύτερο κόπο και προβλήματα τους διερμηνείς. Στην πολύ διεργασία δε μπορούμε να ε, έχουμε υποστηρικτικά μέσα όπως η, η, το να κρατάμε σημειώσεις ή το να κάνουμε κάποια μικρά σχέδια ή συνδέσμους, links όπως λέμε στα αγγλικά. Επίσης μια άλλη ερώτηση, η χρήση της χειρονομίας, οι κινήσεις των χεριών την ώρα που μιλάει ο Δερμηνέας ενισχύει τη δυνατότητά του να ε, επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του. Υπάρχουν σχετικές έρευνες. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ. Συραρπαστική πραγματικά η ερώτησή σας. Δεν έχουμε έρευνες για την νοηματική γλώσσα. Πριν από μία δεκαετία είχε γίνει μία έρευνα που έδειξε ότι οι διερμηνείς από τη νοηματική δεν δείχνουν τις ίδιες γνωσιακές προσαρμογές με τους υπόλοιπους διερμηνείς. Και η ελευθερία που έχουν να χρησιμοποιήσουν ε, τις, ε, τα χέρια τους και να κάνουν χειρονομίες αντί να χρησιμοποιούν το στόμα τους. Φαίνεται ότι ελευθερώνεται το σύστημα το ακουστικό ώστε να είναι πιο ξεκούραστο το έργο τους. Φυσικά είναι έντονο το έργο, αλλά υπάρχει λιγότερη σύγκρουση, οπότε λιγότερη διαχείριση στρες ό,τι αφορά το input και το output. Πάντως δεν υπάρχουν ε, επαρκείς έρευνες για το πώς ε, λειτουργεί ο εγκέφαλος σε περίπτωση νοηματικής διερμηνίας. Πάντως πραγματικά είναι συναρπαστικός και αυτός ο τομέας. Και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις, τις χειρονομίες, η χρήση της κίνησης της χειρονομίας, όχι μόνο για την έκφραση και την κατανόηση, αλλά και για την ε, διατήρηση του, του σήματος, της, του, του νοήματος, για να δείξει κανείς το νόημα. Και πώς επίσης σχεδιάζουμε την εκφορά του λόγου, την ε, ακολουθία και περίπλοκων ε, λέξεων όταν αποδίδουμε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω, ίσως ε, και οι συνάδελφοι θα ήθελαν να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημά σας. Σε ό,τι φορά τις μελέτες, νομίζω ότι έγιναν έρευνες σε σχέση με τα σκαριθήματα που κάνουμε, τα σχέδια που κάνουμε στην καμπίνα μερικές φορές κάνοντας κάτι άλλο, και όντως είναι περίεργο αυτό, φαίνεται ότι ακριβώς επειδή κάνουμε κάτι άλλο ταυτόχρονα, αυτοματοποιούμε κάποιες άλλες ε, ενέργειες. Και όταν ο, ο μιλητής μιλάει πολύ γρήγορα, πολλοί διερμηνείς κλείνουν τα μάτια και αυτό τους βοηθάει στη συγκέντρωση. Βέβαια, ε, ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί 80% των, ε, των πόρων του, αλλά φαίνεται ότι ε, ε, αν ταυτόχρονα κάνουμε κάτι με τα χέρια, γράφουμε κάτι, κάνουμε κάποια σκαρυφήματα, απελευθερώνουμε κάποιους ε, ακουστικούς σπόρους. Χαίρομαι που δεν βλέπει κανένα στις δικές μου μουτζούρες στην καμπίνα. Το όνομά σας. Αλή Τεντσαν από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία και νομίζω ότι εφόσον υπάρχει διερμηνία από τα τουρκικά μπορώ να μιλήσω τουρκικά. Έχω μια ερώτηση για τον ε, καθηγητή Ερβέ Αντελμαν. Εγώ πρώτη φορά βλέπω αυτό που λέτε, αλλά βλέπω ότι ξέρετε πολύ καλά το ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι συναδέλφων που μπορούν από τρεις, τέσσερις, πέντε διαφορετικές γλώσσες να μεταφράζουν. Και μας μιλήσατε για τον ε, κερκοφόρο πυρήνα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν ο κερκοφόρος πυρήνας μπορεί με, την αύξηση των γλωσσών που μαθαίνει κανείς να ενισχυθεί, αν έχετε κάποια τέτοια παρατήρηση. Euh, Σε ευχαριστώ για την ερώτησή σας η οποία είναι πάλι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν είχαμε την δυνατότητα με την ομάδα μου να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει όμως έρευνα η οποία γίνεται για τους πολυγλώσσους, όχι, όχι οι διερμηνείς εννοώ, που αποδεικνύει ότι όσο καλύτερα μιλάμε τις ξένες γλώσσες τόσο λιγότερες συγκρούσεις μεταξύ τους υπάρχουν. Οι διερμηνείς τους οποίους έχουμε εδώ μπροστά που μπορούν με τέτοιο θεαματικό τρόπο να μεταφράζουν τόσες γλώσσες είναι άτομα που ελέγχουν πολύ καλά τις αρχικές τους γλώσσες, τις γλώσσες πηγής δεν έχει σημασία το να έχουν τρεις, πέντε ή έξι γλώσσες στο συνδυασμό τους. Από όλα αυτά υπάρχουν κάποια όρια στον τομέα αποθήκευσης των πληροφοριών των γλωσσικών. Μια γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε λιγότερα στον επαγγελματικό τομέα διότι δεν μας δίδεται η ευκαιρία είναι μερικές φορές πιο δύσκολη στην χρήση της. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ε, ποιοι είναι οι συσχετισμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιες είναι οι δομές οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιούμε μία γλώσσα ε, ε, την οποία δεν ελέγχουμε πάρα πολύ διότι δεν έχουμε ασχοληθεί μαζί της εδώ και ένα χρόνο. Αλλά δυστυχώς άμεσα στην ερώτησή σας δεν δίναμε να απαντήσω. Um, ένα επιπλέον ερώτημα για τους ερευνητές. Ένας εδώ και μετά πιο πίσω. Παρακαλώ το όνομά σας. Σα ε, σας ευχαριστώ λοιπόν. Γκοντσαρέφ λέγομαι από το Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ε, σκεφτεί τους λεγόμενους, ε, τα λεγόμενα νευρώνια καθρέφτες και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσουν την, εκπαίδευση των διερμηνέων. Το μυστικό αυτών των συσχετήσεων ανάμεσα στους μουσικούς και τους διερμηνείς ίσως τελικά και να έγκυται στην ικανότητα την οποία έχουν να εργάζονται μέσω αυτών των νευρονίων καθρεπτών Νομίζω ότι αυτή είναι μια έννοια η οποία έχει ερευνηθεί και η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας στην Ιταλία. Στην Ρωσία έχουμε έναν πολύ γνωστό βιολόγο και γλωσσολόγο, την Τσιτσνιεύσκα, η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό των καθρεπτών νευρονίων. Έχω τώρα και μια συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με αυτό που λέμε στα αγγλικά multitasking. μιλώντας ακριβώς και την ε, δυνατότητα της πολλαπλά επηρεαζόμενης και σχηματιζόμενης σκέψης στα πλαίσια της επεξεργασίας των πηγών. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την διερμηνία, αφορά πάρα πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες και είμαι βέβαιος ότι εδώ θα υπάρχουν πολύ περισσότερες ε, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες θα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μεθόδους. Τώρα, ε, σχετικά με τη μουσική και τις γλώσσες μπορεί κάποιος να βεβαιώνεται για τις ικανότητές του αυτούς τους τομείς από μόνος του. Well, merci. Ε, je... Σας, σας ευχαριστώ. Ό,τι αφορά τους νευρώνες κάτωπτρα, που όντως ανακαλύφθηκαν στην Ιταλία από τον καθηγητή Ριτζολάτη, πραγματικά Πολύ εύστοχη ερώτησή σα. Μια και υπάρχει μεγάλη σύνδεση και διαρθρωτική και λειτουργική μεταξύ της παραγωγής του λόγου και τη κατανόηση του λόγου, φαίνεται ότι ένα τέτοιο νευρονικό δίκτυο που αντανακλά ουσιαστικά αντικατοπτρίζει αυτό που ακούμε στην εκφορά του λόγου μας θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αν αντίθετα ε, θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια χαρτογράφηση άμεση μεταξύ αυτού που ακούμε και της ενεργοποίησης ε, του, του μοντέλου παραγωγής ε, του, της πληροφορίας αυτής, τότε το μοντέλο αναπαραγωγής θα είχε πρόβλημα, γιατί θα έχουμε ουσιαστικά ενεργοποιήσει το σύστημα παραγωγής ε, για τη γλώσσα που ακούμε, τη γλώσσα πηγής. Ως προς τη φωνολογία, ας, ας φανταστούμε ότι ξεκινάει ο διερμηνέας να παράγει την γλώσσα που ακούει, θα έχει όμως πρόβλημα προβλήματα στο, στο τονισμό, στην ε, μελωδικότητα. Και σε ό,τι αφορά την παραγωγή, το τελικό προϊόν θα είναι χρήσιμο. Ε, θα ήταν δύσκολο να περάσει σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ελέγξει ο Δερμηνέας και να καταργήσει, να καταπιέσει, να αποθήσει αυτή την τάση που έχει. Και αυτό το κάνει ο κερκοφόρος πυρήνας που ακριβώς αναστέλει, καταπιέζει κάποιες δράσεις που είναι ακατάλληλες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το σύστημα όμως των νευρώνων κατόπτρων θα μας διδάξει πολλά για το πώς ε, χρησιμοποιούμε την νήμη εργασίας όταν ε, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Κατά τη γνώμη μου εκεί θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τους ε, νευρώνες κάτωπτρα. Ελπίζω να απάντησα τουλάχιστον έστω σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό που παρατηρήσαμε με ενδιαφέρον στη διαδικασία της κατάρτισης των διευμεριών για το πώς αποκτούν τις ε, δεξιότητές τους Μερικές φορές ε, ε, αυτές οι παρεμβολές δεν ε, ανακύπτουν από την αρχή, αλλά κάπου στη μέση της κατάρτισης και είναι δύσκολο να εκριζωθούν. Και σε επίπεδο φωνεμάτων αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκεί έχουμε περισσότερες παρεμβολές και μερικές φορές δεν το συνειδητοποιούν οι ασκούμενοι. Χρειάζεται πολύ εξάσκηση και πρακτική ιδιαίτερα το κουραζόμαστε. Και αν μαγνητοσκοπούσαμε τη διερμηνία μας, θα διαπιστώνουμε ότι όσο περισσότερο κουραζόμαστε, τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να εντοπίζουμε αυτές τις παρεμβολές. Και όλο και περισσότερες τέτοιες παρεμβολές έχουμε. Ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις και σας καίνε, αλλά παρακαλώ ο κάθε ομιλητής που λαμβάνει το λόγο να θέτει μία ερώτηση. Όντως έχω πληθώρα ερωτήσεων. Επικεντρωθείτε σε μία, στην πιο σημαντική. Έχω τρεις. Δεν ξέρω πια να διαλέξω. Αυτά που μάθαμε από τις μελέτες του καθηγητού Άντελμαν μπορούμε να τα μεταφέρουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουν οι τεχνολογίες ε, στις μηχανές που κάνουν αυτό με τη μετάφραση. Μια και ήταν αφηρημένη συντονίστρια, θα επαναλάβω την ερώτησή μου. Αυτά που ακούσαμε από την έρευνά σας μπορούν να μας οδηγήσουν και στην παραγωγή κάποιων ε, ε, μορίων, ε, φαρμάκων για να καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ κάνοντας μια μαγνητική τομογραφία των υποψηφίων για να δούμε τι συμβαίνει στον εγκεφαλό τους. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και με διασκέδασαν πραγματικά. Τώρα απαντώ με αντίστροφη πορεία. Σε ό,τι αφορά τη χρήση της μαγνητικής ε, τομογραφίες για την επιλογή υποψηφίων. Όχι, έχω πολλές επιφυλάξεις ε, και δεοντολογικές. Ακόμη και αν έχουμε τα καλύτερα σκάνερ του κόσμου, που μπορούν να εντοπίσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια του εγκεφάλου, δεν συγκρίνεται κάτι τέτοιο με τη γνώμη του χρήστη, του πελάτη, αυτού που ακούει το προϊόν της διερμηνίας. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε τέτοιες μορφές ε, απεικόνησης μαγνητικής να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα τώρα, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η ερώτηση, γιατί οι ζώνες που ανέφερα στην ε, παρουσίασή μου και σας μίλησα για την όσο του Πάρκινσον, έχουμε πολλές ε, φαρμακευτικές αγωγές που ακριβώς ε, ε, χρησιμοποιούν την τοπαμίνη που είναι πολύ σημαντική για την αυτοπεποίθηση, για την εκμάθηση αλλά κυρίως στις διαδικασίες επιβράβευσης, την, τη συνέστηση ότι κάναμε κάτι καλά. Και υπάρχουν πολλά φάρμακα που δρούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορέσαμε όμως ακόμη να ελέγξουμε την ενέργεια αυτών των φαρμάκων στους δερμηνείς, γιατί αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για όσους ε, είναι ε, ασθενείς με Πάρκινσον. Ακούγονται πολλά στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα smart drugs. Και οι φοιτητέ ε, μπορούν να προμηθεύονται χωρί συνταγογράφηση μέσω του διαδικτύου τέτοιου του φάρμακα που μπορεί να διαταράξουν την ε, συγκέντρωσή τους ή να ενισχύσουν τη συγκέντρωσή τους παροδικά τουλάχιστον, αλλά πραγματικά δεν θα ενθάρρυνα κανέναν να κάνει πειράματα με τέτοια φάρμακα, γιατί αυτά τα smart drugs, αυτά τα έξυπνα ναρκωτικά έχουν ε, πολλές παρενέργειες. Τώρα, για τα μηχανήματα, τι συσκευή δεν νομίζω ότι η έρευνά μου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη τεχνολογίας για τέτοιες συσκευέ αυτόματης μετάφρασης. Εγώ δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό πάντως. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι βρίσκουμε κάποια δίκτυα που ε, αφορούν τον έλεγχο. Αν θέλουμε μια συσκευή λοιπόν που να κάνει μετάφραση όπως ο άνθρωπος, θα πρέπει να έχουμε ε, μία έξοδο του μηνύματος ε, με τρόπο που θα συμβολίζει ακριβώς την αντίστοιχη. Δεν νομίζω ότι καν τα ρομπότ να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια, στο μέλλον κατά τη ε, δημιουργία συστημάτων φαντάζομαι θα παραπέμπουμε σε τέτοιες έρευνες, αλλά πόρο απέχουμε ακόμη από κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Μια σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση ο καθηγητής Σκοπονσκή. Ευχαριστώ. Υπάρχει πιστεύω σημαντική ταύτιση μεταξύ της ακουστικής στη μουσική και της ακουστικής στη γλωσσική επεξεργασία. Ε, θα ήθελα όμως να μου πείτε πώς λειτουργεί αυτό και μια άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Θα καλούσα τους συναδέλφους να σηκώνουν το χέρι τους αν παίζουν κάποιο όργανο μουσικό και αν μπορούν να διαβάσουν παρτιτούρα όταν τραγουδάνε. Πόσοι από εμά μπορούν να το κάνουν αυτό. Ε, και τα δύο, καλά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να προβώ στην εξή παρατήρηση. Αν συγκρίνουμε διαφορετικά ε, μουσικά όργανα, υπάρχουν όργανα όπως το βιολί, όπου η επεξεργασία είναι οριζόντια. Διαβάζουμε την παρτιτούρα από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως διαβάζουμε τις περισσότερε γλώσσες στο αραβικά δεξιά προς ε, αριστερά, αλλά οριζόντια. Ορισμένες άλλες όμως ε, Ορισμένε όμω ασιατικέ γλώσσε δεν διαβάζουν αριστερά-δεξιά-δεξιά-αριστερά, αλλά κατακόρυφα. Και στο εκκλησιαστικό όργανο διαβάζουμε ένα κλειδί στο ένα χέρι και ένα πεντάλι στο ένα πόδι και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη περιπλοκή στην πόλη επεξεργασία. Γι' αυτό λοιπόν θα κατέληγα στο ερώτημα εάν είναι Πεφερυπίνο ή Ιάπωνας που διαβάζει κατακόρυφα καλύτερος πιθανόν στο να παίζει εκκλησιαστικό όργανο από ότι ένας Ευρωπαίος που διαβάζει οριζόντια. Σαν αστείο λίγο πολύ το λέω. Και επίσης ε, η παραγωγή του ήχου είναι διαφορετική ανάλογα με το όργανο. Ε, ορίζεται, ε, το πιάνο έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα ήχου, ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Το βιολί δεν έχει περιορισμένο ηχόχρωμα ή φάσμα ήχου με ελάχιστη ε, διακίνηση των ε, δακτύλων μπορούμε να αλλάξουμε την μουσική που βγάζει. Ξεκινάω εγώ, λέει κυρία ε, Λουαζού, και μετά η Μάγδα. Για την ανάγνωση. Μπορεί, μπορεί για τους Ιάπωνες που λέτε, γιατί όντως το εκκλησιαστικό όργανο είναι αυτό από τα όργανα τα οποία απαιτεί περισσότερες δυνατότητες πολυδιεργασίας, όπως άλλωστε και η Διεύθυνση Ορχήστρας, γι' αυτό όταν κοιτάω όταν μελετάω τους διευθυντές ορχήστρας το διαπιστώνω αυτό. Αλλά η σύγκριση με τον ε, παίκτη, με τον μουσικό του εκκλησιαστικού οργάνου είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ ε, διαργασία. Για τους Ιάπωνες η σύγκριση δεν ξέρω αν μπορεί να ευσταθεί, αλλά πάντως όταν έχουμε πολλά επίπεδα και το, πνευ... και το βλέμμα μας δεν πάει, ε, ας πούμε τα δύο μέτρα που έχουμε, το βλέμμα μας δεν ανεβατεβαίνει από το ένα μέτρο στο άλλο για το πιάνο φερρυπίν δεξιά-αριστερό χέρι, αλλά τα, τα πηγαίνει παράλληλα και αυτό νομίζω ότι ισχύει και για το γραπτό λόγο. Θες να συνεχίσεις. Να μιλήσω ισπανικά. Όντως, πολύ εύστοχο το σχόλιο σας και το έλαβα υπόψη στα μοντέλα που έκανα, γιατί τα μοντέλα για τη μουσική με συνοδεία ένας μουσικός ε, ένας πιανίστας που διαβάζει μια παρτιτούρα διαβάζει τουλάχιστον ε, τρεις σειρές ταυτόχρονα. Ανάλογα με το με πόσους μουσικούς παίζει, αν είναι τρίο ή κουαρτέτο. Ενώ ε, στο εκκλησιαστικό όργανο είναι περισσότερο κάθετη η ανάγνωση. Κάτι που κάνει πιο δύσκολο το, το multitasking, την πολυδιεργασία. Ένας πιανίστας που συνοδεύει πολλούς ε, παίκτες ε, εκκλησιαστικού οργάνου κάνει πραγματικά πολύ διεργασία γιατί διαβάζει ταυτόχρονα αριστερό, δεξιό χέρι, τα πετάλια και προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές όσο προχωράει στην ανάγνωση της παρτιτούρας. Οπότε γίνεται πολύ πιο περίπλοκη, πολύ διεργασία. Multitasking έντονο έχουν και οι διευθυντές ορχήστρας, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, κατά το διάλειμμα του καφέ. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους. Και τώρα πάμε στο πιο δύσκολο εγχείρημα, τη πιο δύσκολη στιγμή του φόρουμ, την αναμνηστική φωτογραφία. Μόλις ήρθε ο φωτογράφος και αν επιδείξουμε πειθαρχία και οργάνωση και βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία αναμνηστική, θα μπορέσουμε να πιούμε και ένα καφέ. Επιστροφή στην αίθουσα σε 10.30 για να ακούσουμε άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ο φωτογράφος θα σας τοποθετήσει που κρίνει απαραίτητο για να βγάλει μια ωραία φωτογραφία. Α, είναι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 Ladies and gentlemen, could you take your seat, please? Please go back. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ. Και βάλτε παρακαλώ ακουστικά αν δεν καταλαβαίνετε γερμανικά, διότι σκοπεύω να μιλήσω γερμανικά για να σας παρουσιάσω την επόμενη ομιλήτρια και συνεχίσω να μιλάω όσο να φορέσετε όλοι τα ακουστικά σας και να βρείτε και το κανάλι της διερμηνίας γιατί θέλω να μιλήσω γερμανικά καλωσορίζοντας τη νέα ε, προσκεκλημένη με την επόμενη ομιλήτριά μας, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά γερμανικά και επίσης θα θέλω να πω κάτι πολύ σπάνιο, έχει ως μητρική γλώσσα την Ιρλανδική, μαζί με τα Αγγλικά, είναι διευθύντρια του Lingua Center, Language Center, γλωσσικού κέντρου στο, στην Ιρλανδία έχει βέβαια την εμπειρία στη δασκαλία των γλωσσών, αλλά ιδιαίτερα έχει αγωνιστεί για την προαγωγή της Ιρλανδικής γλώσσας. Εργάζεται στο Ιρλανδόφωνο ραδιόφωνο και γενικά βοηθάει στην προώθηση της χρήσης της γλώσσας. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Language Testers Europe. Καθηγήτρια Γκάλαχερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Σουζάνε. Αρχίζει, αρχίζει κελτικά η κυρία Κάλαχερ. En seo a loirt ar náhairta ar náhar show a seo agus bhil mar ráfasta bhfuil más mór agam er obair na Parliamente Maidir le corthaí. Συνεχίζει κελτικά η κυρία Γκάλαχερ. Ε, μάσκ, τσάνκα, Euh, Θα ξεκινήσω με κάποιους ε, ορισμούς. Κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα σε δύο μορφές πολυγλωσσίας. Λοιπόν, από τη μία έχουμε τη συμβίωση διαφορετικών γλωσσών σε μία δεδομένη κοινωνία ενώ αντίθετα η άλλη πολυγλωσία αναφέρεται ε, στις αποσκευές της γλωσσικές του συγκεκριμένου προσώπου κάθε φορά σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης την οποία θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Λίγκουα φράγκα και εδώ έχουμε διαφορετικού τύπου ορισμούς. Χρησιμοποιώ τον όρο ε, ως βοηθητική γλώσσα σχέσεων που χρησιμοποιείται από ομάδες που έχουν διαφορετικού τύπου μητρικές γλώσσες, διαφορετικές μητρικές γλώσσες. Είναι μια ενδιάμεση δηλαδή γλώσσα. Την 1η Ιανουαρίου του 1973 η Ιρλανδία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και οι αντίθετοι με αυτό το ιστορικό συμβάν θεώρησαν ότι δεν είχε και καμιά άλλη επιλογή γιατί ακολουθούσε υποχρεωτικά το Ηνωμένο Βασίλειο από το οποίο έχει εξαρτηθεί η οικονομία της αλλά η πλειοψηφία ήταν υπέρ. Έβλεπε ότι υπάρχει ένα νέο μέλλον πέραν των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, πέραν από την απεικιοκρατία, ένα μέλλον που θα καθιστούσε την περιοχή πιο πλούσια, πιο περίπλοκη και πιο ευρωπαϊκή. Για να πάρει κανείς πλήρες, ε, να, να παίξει <clears throat> τον ρόλο πλήρους μέλους έπρεπε να μάθουμε κάποιες ξένες γλώσσες, κυρίως τα γαλλικά και τα γερμανικά. Αυτό πήρε κάποια χρόνια αρχίσαμε να διαβάζουμε για το Μοπασάν στο σχολείο όπως το κάναμε παλιότερα και με τον Τίτο Λίβιο. Παρ' όλα αυτά το όραμα μιας πολυγλωσσικής Ευρώπης και ο ρόλος της Ιρλανδίας σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι το οποίο άρχισε σιγά σιγά να μην είναι μπροστά μας. Παρά διάφορα συνέδρια και συναντήσεις που είχαν σαν θέμα ότι τα αγγλικά μόνα τους δεν <clears throat> αρκούν, η πολυγλωσία κατέστη ένα, μια παράλληλη πραγματικότητα και μάλιστα σε μια γλώσσα που αναγνωρίζει δύο επίσημες γλώσσες στο σύνταγμά της, σε μια χώρα συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε στην αρχή της ενότητας στη διαφορετικότητα. Από τις αρχές της η γλωσσική της πολιτική είχε σαν φιλοδοξία να ενθαρρύνει τους πολίτες των κρατών μελών να μάθουν δύο ή τρεις άλλες γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλιότερα κοινότητας, παλιότερα αγοράς, έτσι ώστε και για οικονομικούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους να επιτραπεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία μακροπρόθεσμα ε, ή μάλλον ο στόχος ο μακροπρόθεσμος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες των πολιτών έτσι ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες εκτός της μητρικής. Ο ορισμός αυτού του στόχου διαφεύγει από πολλούς από τους συμπολίτες μας σήμερα. Ε, όρος μητρική γλώσσα είναι όρος βεβαρημένος. Οι Ιρλανδοί αγγλόφωνοι σαν παράδειγμα ομιλούν για την επιθυμία τους να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, αναφερόμενη στα κελτικά, την οποία μερικές φορές ονομάζουμε γοηδελικά και πολλοί από αυτούς δεν ελέγχουν ουσιαστικά. Ταυτόχρονα ο όρος αυτός, μητρική γλώσσα, χρησιμοποιείται στον ενικό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινότητα μονογλωσσικών εθνών. Στην τελική έκθεση του προγράμματος βαλέρ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Τζοάννα Μακπέκ ε, δίνει έναν καλό ορισμό. Λέει ότι χαρακτηρίζουμε τις πολιτικές του τέλους του 20ου αιώνα μονογλωσσικές, διότι στην ουσία ε, προτείνουν ότι ο καθένας έχει μια πρώτη μητρική γλώσσα και ότι όλοι θα αποκτήσουν μια δεύτερη γλώσσα στη συνέχεια. Με παρόμοιο τρόπο, με έναν τρόπο διδακτικό τυπικά συγκρίσιμο. Θεωρούμε ότι οι δύο άλλες γλώσσες σημαίνει δύο γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τι γίνεται σε περιπτώσεις όπως η Ιρλανδία και κάποιες άλλες χώρες που εκπροσωπείται εδώ σήμερα που έχουν πάνω της μία επίσημης γλώσσας ή αυτές που έχουν μειονοτικές γλώσσες που δεν αναγνωρίζονται επίσημες γλώσσες ή γλώσσες εργασίας. Η έκθεση Ευρυδίκη του 12 για τη διδασκαλία των γλωσσών στα σχολεία δείχνει ότι πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Η επίσημη Ευρώπη τώρα. Ο Γκάουκ θα ήθελε να μιλάει αγγλικά η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τις υποθέσεις σε τρεις διαδικαστικές γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Μετά από την διεύρυνση προς Ανατολά στο 4, η χρήση των γαλλικών στις συνεδριάσεις μειώθηκε και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο ρόλος της γερμανικής σαν διαδικαστική γλώσσα δεν υπάρχει παρά μόνο στα χαρτιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τώρα 24 επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας κατά συνέπεια, Ακούμε όλο και περισσότερες αρνητικές, ε, αρνητικά σχόλια γύρω από τη μετάφραση που έχει κόστος ένα δις <clears throat> τον χρόνο, δηλαδή όπως λέει κάποιος ένα ποτήρι καφέ, μια κούπα καφέ τον χρόνο για κάθε πολίτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι με, τα, την κατάσταση που ισχύει σήμερα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες. Πέρυσι πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου της προεδρίας του ο Γιώαχιμ Γκάουκ, ο Γερμανός Πρόεδρος, είπε ότι θα πρέπει να έχει μια κοινή γλώσσα και αυτή η γλώσσα θα έπρεπε να είναι τα αγγλικά και μας είπε τα εξής στα γερμανικά. Περισσότερη Ευρώπα δεν σημαίνει περισσότερη πολυγλωσία για τις ελίτ, αλλά πολυγλωσία για μεγαλύτερες ακόμη ομάδες πολιτών, για περισσότερους διαρκώς ανθρώπους και τελικά για όλους. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούν και τα δύο να συνεπάρξουν στην Ευρώπη και η ενύπαρξη μέσα στην μετρική γλώσσα και την ποιησή της, αλλά και μια πρακτικά χρήσιμη αγγλική γλώσσα για κάθε μορφή ε, βίου, κοινού βίου και κάθε ηλικία και συνεχίζει το όραμά του. Με μια κοινή γλώσσα συνεχίζω το όραμά μου για μια μελλοντική Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή αγορά, ένα κοινό χώρο συζητήσεων για την, για την ε, ανταλλαγή δημοκρατικά των απόψεων και των θέσεων. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, Μπορεί το όραμα του Προέδρου Γκάουκ να πραγματοποιείται τελικά, αν και κατά τρόπο παράδοξο ο αριθμός των Βρετανών που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ριζικά μειωθεί, αποτελούν δηλαδή το 86% του εκτελεστικού προσ... το 4,6% του εκτελεστικού προσωπικού, πολύ χαμηλότερο από το 2,5% που είναι το ποσοστό του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν οι κάτοικοι της χώρας αυτή. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη όσον αφορά την αναλογία Ιρλανδών που ε, ε, εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ε, επιβεβαιώνει δόθηκε πρόσφατα από έναν ανώτερο Ευρωπαίο υπάλληλο στο ε, Δουβλίνο, ο οποίος ε, ε, σχολίαζε ηρωνικά την υποβάθμιση του αριθμού των αγγλοφώνων ο πρόεδρος Γκάουκ μπορεί να έχει πολύ καλές προθέσεις, ωστόσο θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το όραμά του για την αγγλική αλλά και για τις άλλες γλώσσες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αντιστοιχεί απολύτως στην διγλωσία, όπως την έχει επαναδιατυπώσει ο Φίσμαν. δηλαδή τη συνύπαρξη δύο γλωσσών ή δύο εκδοχών γλώσσας, δίπλα-δίπλα μία στην άλλη, όπου η πιο ε, υψηλού επίπεδου, εν προκειμένου η αγγλική χρησιμοποιείται στις τυπικές ε, και επίσημες ευκαιρίες και εκδηλώσει, ενώ η δεύτερη, η λιγότερο ε, αποδεκτή, με λιγότερο κύρος, χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Και έτσι μπορεί να αναφέρεται διαρκώς η διεύρυνση προς ανατόλα του 2004 ως ο κινητήριος μοχλός για την ηγεμονία της Αγγλικής στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και αν αυτή η εξέλιξη υπέρ της Αγγλικής έχει πηγή τις πολιτικές, τις γλωσσικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ε, αυτές που προσπαθούν να επηρεάσουν την εκμάθηση και την απόκτηση ξένων γλωσσών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη έχει γίνει σε σχέση με τις πολιτικές ε, και τις στρατηγικές για τη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Βόντακ και Κριανιόφσκι, που μιλούν για μια εντυνόμενη γλωσσική ε, χρηστικότητα με υπόβαθρο την οικονομία που στηρίζεται στη γνώση, όπου οι γλώσσες θεωρούνται μόνο δεξιότητες. Από το 2008 ωστόσο βλέπουμε ότι ξαναγυρνάμε στα οικονομικά επιχειρήματα και πάλι με τους δύο αυτούς ερευνητές οι οποίοι μας λένε φαίνεται προφανές πως ε, οι πολιτική για τις γλώσσες και την πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, αποκτήσει, έχει προσκτήσει μεγαλύτερη και ευρύτερη κατανόηση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού ρόλου των γλωσσών και της πολυγλωσσίας και δυστυχώς αρχές ε, της οικονομικής κρίσης το 2008 και λόγω της μεταφοράς του χαρτοφυλακίου πολυγλωσσίας στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χαρτοφυλάκιο πολιτισμού εκπαίδευσης και νεολαίας του 2010. Πολλές από τις πολιτικές αυτές του 2008 δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και έτσι οι πολιτικές με βάση τις ε, προοπτικές Λισαβόνας δεν έχουν υλοποιηθεί. Τέλος παραθεστώ, Σεπτέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ένα ανακοινωθέν με τίτλο χώρο συζητήσεως των θεμάτων που αφορούν τις γλώσσες στην Ευρώπη με τη μορφή ερωτηματολογίων και ε, την απασχολεί αυτή την ανακοίνωση η δυνατότητα της αγωγής μιας ενιαίας γλώσσας. Η απάντηση είναι εξή. Παρά είναι απλουστευτικό το να θεωρούμε ότι μια ενιαία γλώσσα μπορεί να, σε όλες, να ανταποκριθεί σε όλες τις γλωσσικές ανάγκες. αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα δίνει έμφαση στην ε, ποικιλία και όχι στην ομοιομορφία σε σχέση με την πολυγλωσσία. Αυτή η δήλωση είναι καθησυχαστική, ωστόσο η πραγματικότητα φαίνεται να φαίνεται να απορρίπτει αυτή τη δήλωση, να τη διαψεύδει, γιατί βλέπουμε ότι ο στόχος ε, βέβαια μπορεί να είναι πολύ καλός και άξιος, αλλά ταυτόχρονα και δαπανηρός το να έχουμε δηλαδή πολλές γλώσσες. Η πολύγλωση Ευρώπη, η πραγματικότητα ε, στην Ευρώπη, η πραγματικότητα στην πράξη στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική. Η Ευρώπη, δεν έχει ποτέ υπάρξει τόσο πολύ γλώσσα. Στο Ευρωπαϊκό Ευρωβαρόμικρο του 2012 έχουμε 23 αναγνωρισμένε γλώσσες, τώρα είναι 24, με πάνω από 60 τοπικές μειονοτικές περιφερειακές γλώσσες και μεγάλο αριθμό μη τοπικών γλωσσών που ε, χρησιμοποιούν οι κοινότητες των μεταναστών. Το 2007 το έργο Valor που ήδη αναφέρθηκε νωρίτερα κατέγραφε 440 γλώσσες ομιλούμενες και τουλάχιστον 18 νοηματικές γλώσσες στις 21 χώρες που συμμετέσχουν στην έρευνα. Στην Ιρλανδία το 2005 οι δικές μας έρευνες αποκαλύψαν την ύπαρξη τουλάχιστον περίπου 200 γλωσσών που ομιλούνται ή χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Ιρλανδία, μια χώρα που έχει λίγο περισσότερο από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ένα σύνολο 167 ε, καταγεγραμμένων γλωσσών δεν ελάμβανε σε προηγούμενη περίοδο υπόψη αριθμό βιονοτικών γλωσσών όπως το Κασούμπ, γιατί αυτές δεν καταγράφονταν στα διοικητικά έντυπα ή στα αιτήματα για μετάφραση όταν, χρησιμο... όταν ζητούσε κάτι τέτοιο ένας ε, ξένος ομιλητής που χρησιμοποιούσε δηλαδή την ε, γλώσσα της πλειοψηφίας. Παρά τη σημαντική οικονομική ύφεση, η Ιρλανδία διατηρεί πολύ σημαντικό ποσοστό πολυγλωσσίας με 182 γλώσσες στην απογραφή του 2011 και 26% των ομιλητών ξένων γλωσσών που έχουν γεννηθεί στην Ιρλανδία. Και σας παραθέτω, στην περίπτωση των ε, αλλοδαπών ευρωπαϊκής καταγωγής πρώτη γλώσσα είναι τα πολωνικά και τα ακολουθούν η λιθουανική, η ρωσική, η ρωμανική και η, Λατβ... λετωνική γλώσσα, ενώ οι προερχόμενοι από την Ασία μιλούν ε, φιλιπ φιλιππίνο, κινέζικα, μανταρίν και Καντονή, μαλάι, ουρντού και χίντι. Ιδέα Αφρικανική πρόέλευση. Κυρίω έχουν την Ιωρούμπα, μετά έχουν γαλλικά, αφρικανικά και Αφρικάν. Και στην Βόρεια και Νότια Αμερική, Πορτογαλικά κυρίω και μετά Ισπανικά, Γαλλικά, Πολωνικά και Γερμανικά. Και στο παράδειγμα αυτό είναι πολύ πιθανό οι 182 γλώσσε που αναφέραμε να μην είναι η ακριβή εκτίμηση, γιατί κατά την εμπειρία μα, κατά την πείρα μα, οι απόδημοι μετανάστες ε, ελεγχιστοποιούν τον αριθμό των γλωσσών που γνωρίζουν. Αυτό συμβαίνει κυρίως στους Αφρικανούς που αδιαφορούν για τις γλώσσες που δεν είναι γραπτές. Και συνήθως ε, για την ε, ερώτηση που τους θέτε είναι μιλάτε άλλη γλώσσα πριν των Αγγλικών ή των Ιρλανδικών στο σπίτι. Ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να ερμηνεύσουν κατά γράμμα την ερώτηση αναφερόμενοι σε μία μονογλώσσα, ενώ στην ουσία μιλούσαν πολύ περισσότερες. Ε, μάλιστα είδαμε και γνωρίσαμε και από, ε, μετανάστες στην Ιρλανδία που ακριβώς το γεγονός ότι συμμετέχουν σε μία πολύγλωση κοινότητα τους ενοχλεί γιατί είναι πεπισμένοι ότι μία μόνο γλωσσική παράδοση έχει περισσότερο κύρος. Σίγουρα αυτό είναι ένα κατάλοιπο ενός απεικιοκρατικού βιώματος. Τώρα, οι μειονότητες ε, που έχουν μια νοοτροπία περισσότερο μονογλωσσική. Ο Γάλλος γλωσσολόγος Αλεξάνδρε Φρανσουά συνοψίζει πολύ καλά την καθημερινότητα πολλών ε, χρηστών μειονοτικών γλωσσών. Οι, ε, οι γλωσσικές μειονότητες υφίστανται συνεχώς πιέσεις να απεμπολίσουν τη χρήση της γλώσσας τους και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα της πλειονοτικής ομάδας. Και μάλιστα συνήθως συνδέεται αυτή η πίεση με οικονομική, σχολική, κοινωνική και μια τάση για μια ομοιομορφοποίηση γλωσσική. Έχουμε λοιπόν ιδεολογίες σχεδόν αμυγός μόνο γλωσσικές που ε, χάρη τη συνοχή μιλούν για τη χρήση από όλους μιας ενιαίας γλώσσας. Ε, κατά το, το μοντέλο των Ιακωβίνων που έχει μεγαλύτερα στη Γαλλία, στην Κίνα και αλλού, οι ε, γλωσσικές μειονότητες θεωρούνται ως παράγοντας διαίρεσης. Αγνοούμε, ξεχνάμε πολύ γρήγορα ότι ο, άνθρωπος είναι ικανός να μιλήσει πολλές γλώσσες. Για παράδειγμα, στο, στο ο αγγλόφωνος ο μονογλωσσισμός είναι πολύ περιορισμένος ε, και δεν εκτίθενται οι αγγλόφωνοι σε άλλες ε, ε λογοτεχνίες. Για παράδειγμα, ε, κατά τη γνώμη της Λοράς Μαρή, που γράφει στο Νοβέλο Observateur, μόνο 1% των ε, πληθυστορημάτων που εκδίδονται στις, κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφράζονται στα γαλλικά. Ε, και ενώ η γλώσσα που κατεξοχή μεταφράζεται στον κόσμο είναι τα αγγλικά, ενώ το 33% των μυθιστορημάτων που διαβάζονται στη Γαλλία είναι μεταφράσεις. Ε, οι μεταφράσεις είναι μόνο 4,5% του συνόλου της συνολικής λογοτεχνικής παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και όλος παραδόξως στην Πολωνία το 46% όλων των βιβλίων που έχουν εκδοθεί είναι μεταφράσεις. Στη Γερμανία το ποσοστό αυτό είναι 12%, στην Ισπανία γύρω στο 24% και στη Γαλλία γύρω στο 15%. Άλλο παράδειγμα, οι αγγλόφωνοι γενικώ είναι κατά της, ε, των, υποτίτλων ε, και γι' αυτό δεν γνωρίζουν μία αγγλόφωνο κινηματογράφο. Και μάλιστα ε, στο ραδιόφωνο κάποιοι διαγωνισμοί τραγουδιού ταινιών που είναι εξορισμού επιφανειακοί περιορίζονται κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο. Ποιος σας κατηγορούσε όμως και στο, στην εκπαίδευση κυριαρχεί η Αγγλοφωνία. Μόνο 6% από τα 50 πανεπιστήμια κύριο στον κόσμο βρίσκονται σε μη αγγλόφωνες χώρες, όπως ε, λέει το Times Higher World University Rankings, που κάνει την αξιολόγηση των ε, κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο για το 2013 και 2014. Κανένα ε, γαλλικό ή γερμανικό πανεπιστήμιο δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κατάλογο με τα κορυφαία πανεπιστήμια. Επίσης ε, και στην ταξινόμηση της Σανγκάης μόνο 8 έχουμε από τις 8 ε, σημαντικότερα πανεπιστήμια που είναι μια αγγλόφωνα, δύο γαλλικά και ένα γερμανικό. Σε πολλές χώρες ε, τα πανεπιστήμια συστήνουν επιτροπές για να βελτιώσουν την καλύτερη εμφάνισή τους σε τέτοιους καταλόγους αξιολόγησης, που είναι πολύ σημαντικό για να προσελκύσουν φοιτητές. Επίσης ε, ενθαρρύνονται εκδόσεις ε, σε χώρες ε, σε άλλες γλώσσες πλην των αγγλικών. Και αυτός είναι ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αυτή. Βέβαια, στα όρια που μας επιβάλλει η αντίληψη του κόσμου υπό μονογλωσσική σκοπιά έχουμε και άλλε συνέπειε, Δύο αγγλόφωνε χώρε, χώρες, Ιρλανδία και η Σκοτία, είναι οι μόνε χώρε τη Ευρώπη, όπου η εκμάθηση μια ε, ξένης γλώσσα δεν είναι υποχρεωτική. Στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία η εκμάθηση γλωσσών είναι υποχρεωτική, αλλά μόνο μέχρι την ηλικία των 14 ετών. Στην ανώτατη, η ανώτερη ανώτατη εκπαίδευση η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλύτερη. Έχουμε όλο και περισσότερα ε, προγράμματα γλωσσών, ακόμη και για ειδικού, αλλά μέσω των Αγγλικών. Οπότε έχουμε ε, ένα μόνο μάθημα στη γλώσσα στόχο, αλλά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, λογοτεχνία, πολιτισμός κτλ. γίνεται κυρίως στα γαλλικά. Ε, Ω εκ τούτου, οι αγγλόφωνοι φοιτητέ που περνούν τα χρόνια με βάση την υποτροφία έρασμο στην υπόλοιπη επιρωτική Ευρώπη δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών. Εκτός κι αν ακολουθήσουν αμυγός αγγλόφωνα προγράμματα. Η κοινή γλώσσα, το lingua franca μεταξύ των φοιτητών έρασμος είναι σχεδόν αποκλειστικά τα αγγλικά. Ας μην ξεχνούμε και φυσικά μία παραμονή ενός χρόνου στο εξωτερικό δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Φυσικά και έχει, και τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις επίκτητες γλωσσικές ε, δεξιότητες στα πρόγραμμα του Έρασμος είναι αρκετά απογοητευτικά και που υστερούν σε σχέση με αυτά που θα περιμέναμε. Είναι γνωστές άλλες και κοινωνικές συνέπειες. Τώρα, το οικονομικό κόστος ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητές τους στις αγγλόφωνες χώρες τα πανεπιστήμια δεν παράγουν διπλωματούχους σε ξένες γλώσσες όπως θα τους χρειαζόταν η αγορά εργασίας. Εδώ και χρόνια στο Δουβλίνο έχουμε τα αρχηγεία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η Google, η IBM, το Facebook και έχουν θέσεις για πολύγλωσσους και χρειάζονται πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως ένας μεγάλος αριθμός νέων Ιρλανδών που θα μπορούσαν να δουλέψουν εκεί φεύγουν από τη χώρα και αναζητούν δουλειά σε άλλες αγγλόφωνες χώρες λόγω ακριβώς της έλλειψης γνώσεων. Το θέμα των γλωσσών είναι ένας από τους παράγοντες, αλλά όχι ο μόνος, που εμποδίζει τους αγγλόφωνους υποψήφιους να πάρουν υψηλές θέσεις στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως είπαμε. Πέρα από το προσωπικό και κοινωνικό κόστος της μετανάστευσης, αυτό το γλωσσικό έλλειμμα των αγγλόφωνων χωρών έχει και διαφορετικού τύπου κόστη. Η Ντάιντρε Hunt καθηγήτρια management στο Πανεπιστήμιο του Κόρκο, σε ένα άρθρο το οποίο λέγεται «Οι γλώσσες και η οικονομία». Μας θυμίζει ότι το 75% του πληθυσμού του κόσμου δεν ομιλεί την αγγλική και το 94% δεν τον ομιλεί σαν μητρική γλώσσα. Οι ανακοινώσεις τύπου για τις γλώσσες στην Ευρώπη, οι οποίες εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2013, επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέει η Χάντ. Τα αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα, η πιο διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κάποιες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ακόμα σήμερα το τμήμα του πληθυσμού της Ένωσης που ε, ελέγχει και γνωρίζει επαρκώς την γλώσσα αυτή και το οποίο δεν ξεπερνάει το 50%. Η καθηγήτρια Χάντ αναφέρεται επίσης και σε μία μελέτη την οποία ε, είχαν κάνει οι Φράνκελ και Ρόουζ που ποσοστικοποίησαν τις επιπτώσεις της έλλειψης γλωσσικών γνώσεων στις επιδόσεις των επιχειρήσεων έδειξαν ότι το κόστος των γλωσσικών εμποδίων ήταν 15 με 22% σε σχέση με τα δασμολογικά τέλη. Ε, εκτιμούν επίσης ότι ε, μια κοινή γλώσσα μπορεί να αυξήσει τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες από 75 με 170%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία των γλωσσών για τις επιχειρήσεις. Το 2006 έγινε μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αξιολογηθεί το κόστος του γλωσσικού ελλείμματος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι κάθε χρόνο χιλιάδες από τις επιχειρήσεις αυτές χάνουν κάποια συμβόλαια λόγω των γλωσσικών μειο... μειονεκτικών καταστάσεων τους. Το 11% των μικρομεσαίων που εξάγουν και που είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο ε, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας. Στην Ιρλανδία έχουν επανειλημμένα οι βιομήχανοι και ο τομέας της τεχνολογίας και της πληροφορίας μεγαλύτερες ε, ε, γνώσεις γλωσσικές, αλλά αυτό δεν έχει αποδώσει τίποτα, δεν ξέρουμε γιατί. Όπως γνωρίζουν όλοι η διδασκαλία των γλωσσών κοστίζει, αλλά η δυνατότητα κατάρτισης των ομιλητών είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Ίσως οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται, αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, δεν πρέπει να καλυφθούν οικονομικά. Πρέπει επίσης <clears throat> να δούμε τι γίνεται στην υπηρετική Ευρώπη. Η εκμάθηση των γλωσσών σημαίνει ουσιαστικά την εκμάθηση των αγγλικών. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα που διδάσκεται περισσότερο σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση Ευρυδίκη, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, το 90% των μαθητών τουλάχιστον μαθαίνουν τα αγγλικά στο επίπεδο SIT 2 και συτ 3 σε επίπεδο δηλαδή ε, ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να πούμε ότι το 2009-2010 το 60,8% των μαθητών της ε, δευτεροβάθμιας μάθαινε δύο γλώσσες. Αυτό δείχνει ότι έχει υπάρξει μια αύξηση 14,1% συγκρίνοντας με το 2004-5. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τα επίπεδα επιτυχίας της διαδικασίας εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας εκτός της αγγλικής. Η μελέτη Survey Lang, η οποία αξιολόγησε τις ικανότητες των μαθητών, προφορική γνώση, γραπτή γνώση και γραπτή παραγωγή των ξένων γλωσσών, είχε σαν στόχο να δώσει την δυνατότητα σύγκρισης των χωρών οι οποίες συμμετείχαν στον τομέα της διδασκαλίας των γλωσσών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κάποιοι δείκτες ε, γλωσσικών ικανοτήτων. ή συμμετέχοντες έδωσαν στοιχεία και για, το πρώτο, ε, για την πρώτη τάξη της ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τη δεύτερη τάξη. Πέρασαν τα τέστα σε δύο ξένες γλώσσες, ε, σε, ανάμεσα στα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, που ερχόντουσαν από 14 ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ισπανία, Εστονία, Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, κάτω χώρες Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σουηδία. Τα αγγλικά ήταν η πρώτη ξένη γλώσσα όλων των χωρών εκτός από το Βέλγιο που ήταν τα γαλλικά. Τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων εντάχθηκαν στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, το ΣΕΡΚΛ. Κάποια αποτελέσματα τώρα. Ας δούμε πρώτα τις χώρες στις οποίες οι μαθητές πήγαν καλύτερα στην πρώτη ξένη γλώσσα, δηλαδή είχαν τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στο επίπεδο Β κεφαλαίο, ανεξάρτητοι χρήστες μιλάμε, για μεμονωμένα πρόσωπα δηλαδή, βλέπουμε ότι η επιτυχία τους κυμαίνεται από 60 μέχρι 81%. Ε, Εστονία, Μάλτα, κάτω χώρες και Σουηδία ήταν οι πιο επιτυχείς. Ας δούμε τώρα και τις αρμοδιότητες, τις ικανότητες σε σχέση με τη δεύτερη ξένη γλώσσα πηγαίνουν από 2, από, συγγνώμη, διορθώνει η ομιλήτρια από 24% σε 60%. Ε, είναι περίεργο που μερικές φορές ε, πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα στα αγγλικά από ό,τι στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Η Γερμανία μάλιστα δεν πήρε μέρος σε αυτή τη μελέτη για... Ιστορικά η Μάλτα συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Η Εσθονία όπου τα ρωσικά ήταν υποχρεωτική δεύτερη γλώσσα δεν είχε τέτοιου είδους συσχετισμούς αν και τα εσθονικά έχουν δανειστεί πολλά από τα γερμανικά στη διάρκεια των αιώνων. Όμως μπορούμε να πούμε ότι επί τη βάση των αποτελεσμάτων του Surveylang οι μαθητές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες μαθαίνουν καλύτερα τα αγγλικά από ό,τι τις άλλες γλώσσες. Η ομάδα του Surveylang καταλήγει στα εξή αποτελέσματα. στα εκπαιδευτικά συστήματα, ακόμα και σε αυτά όπου τα αγγλικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα, οι επιδόσεις στην αγγλική είναι καλύτερες από ό,τι στις υπόλοιπες γλώσσες που ελέγχθηκαν. Αυτό δίνει περαιτέρω αποδείξεις για το ειδικό καθεστώς της αγγλικής γλώσσας και στα ερωτηματολόγια φαίνεται αυτό σχετικά με την αντίληψη που υπάρχει για τη χρησιμότητά της και την δυνατότητα χρήση της στα παραδοσιακά και νέα μέσα. Τέλος παράθεσης. Έχουμε λοιπόν το εξής θέμα στην Ευρώπη, ότι το κύρος της αγγλικής αυξάνεται μαζί με, το, με τη χρήση της και αυτό μπορεί για ορισμένους να θεωρείται ανησυχητικό. Από την άλλη, το καθεστώς γλωσσών άλλων από την αγγλική, ε, τοπικές, εθνικές, ε, περιφερειακές, μειονοτικές γλώσσες ε, σημαίνουν αμφισβήτηση σχεδόν καθημερινή. Ένα καθεστώς ανάμεικτο οδηγεί και σε ικανότητες, δεξιότητες περιορισμένες. Η πολυγλωσία είναι σημαντικός πόρος, σημαντικής αξίας πόρος, που δεν μπορούμε πάντοτε όμω να ποσοστοποιήσουμε την αξία αυτή. Ο αυστραλό, γλωσσολόγο Ζολεμπιάνκο εντοπίζει δέκα διαστάσει τη πολυγλωσία ω πόρου, πνευματική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ή θα γίνει σε σχέση με τη σχέση του πολίτη, δηλαδή με την ε, καταγωγή του δικαιώματα των ανθρώπων του ανθρώπου και θεωρεί ότι η κοινότητα, ένα έθνος ή ένα σύνολο ε, που επενδύει σε όλες τις γλώσσες, ε, κερδίζει ένα καλύτερο επίπεδο, δραστηριότητες περισσότερες, ε, βελτίωση των εμπορικών δυνατοτήτων, βελτίωση των δυνατοτήτων για συμμετοχή σε μια οικονομία της γνώσης, βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, βελτίωση της συμμετοχής στο δημόσιο βίο και τις πρακτικές της δημοκρατίας και καλύτερες στρατηγικές για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, την προώθηση της Τη διαλλακτικότητας, τη ανοχή για τον άλλον και τη αμοιβαία κατανόηση. Άρα λοιπόν για να ολοκληρώσουμε είναι προφανέ ότι ο ρόλος Αγγλική στην Ευρώπη, στην επίσημη Ευρώπη θα ενισχύεται διαρκώ. Δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την πλημμυρίδα, ωστόσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τι άλλε γλώσσε Ευρώπη, ώστε να μην πληγούν από και να μην χάσουν από το, τη θέση τους από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε μια Ευρώπη πολύγλωση που θα δίνει την ίδια αξία σε όλες τις γλώσσες της. Εδώ δεν ε, πρόκειται να θέσουμε ένα τέρμα στη χρήση της Βρετανικής ούτε να παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη μιας lingua franca. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε τα, τα όρια αυτής της lingua franca. Χρειάζεται μια, μια πολιτική στην Ευρώπη, μια πολιτική των γλωσσών που θα προωθεί και θα δίνει αξία σε όλες τις παρούσες γλώσσες που θα αναπτύσσει το δυναμικό του στο γλωσσικό προ όφελο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό κάθε πολίτη τη Ένωσης και ταυτόχρονα θα πρέπει να περιοριστεί η σχέση εξάρτησης μεταξύ αγγλοφώνων και λοιπόν. Όπως κατέγραφε ένας χρονογράφος ε, πέρυσι, καμιά χώρα δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συνθλιβεί από έναν, ομοιογενή τροχό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν τι λένε οι νόμοι αυτό. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να καταλαβαίνουν ποια είναι η τελική εκδοχή του νόμου, αλλά και ε, οι συζητήσει που οδηγούν σε αυτού του νόμου. Αυτό λοιπόν που σημαίνει μεγάλε και γενναιόδορε κινήσει και χειρονομίε προ μικρέ χώρε, Φερρυπίν Μάλτα έχει ίση ψήφο με την Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημαίνει ταυτόχρονα και ενθάρρυνση τη πολυγλωσία και τη ευρυγλωσία, ώστε ε, αυτή να σημαίνει όχι μόνο καλές στα αγγλικά αλλά και, την, ε, και έναν ε, λογικό τρόπο ε, αξιοποίησης όλων των γλωσσών και των κράτων. Σε μια συζήτηση στο Ινστιτούτο Γκέτο το 2006 με τον Γκέρχαρτ Στρίκερ που είναι ο Διευθυντή του Ινστιτούτου γερμανική γλώσσα, που τον, τον ρώτησα να μου προβλέψει ποιο θα είναι το μέλλον των γλωσσών στην Ευρώπη μου λέει και θεωρώ ότι δεν ήταν κωμικό αυτό που μου είπε στα αγγλικά η παράθεση και ζητώ συγγνώμη προ τον καθηγητή Στίκελ η ε, απάντηση λοιπόν ήταν η εξή. Απεσιόδοξο σενάριο. Τα επόμενα χρόνια η εκμάθηση των γλωσσών θα περιορίζεται κατά κύριο λόγο στα αγγλικά. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το ενδιαφέρον προ άλλε γλώσσε ε, θα αρχίσει να μειώνεται ακόμη και για αυτούς που έχουν τις γλώσσες ως μητρικές γλώσσες, τελική, γερμανική, ολλανδική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες εξακολουθήσουν να ομιλούνται αλλά μόνο μέσα στην οικογένεια την ώρα ή την ώρα παίζει κανείς ε, χαρτιά ή που βγαίνει σε μια λαϊκή αγορά. Ενώ τα σημαντικά ζητήματα του κόσμου και τα επαγγελματικά θα ε, λειτουργούν ε, στην επιστήμη και την πολιτική κυρίως με τα ανάμεικτα αγγλικά, τα κρεόλα αγγλικά, αμερικανοαγγλικά, με κάποια στοιχεία γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Στις δε βρετανικές νήσους η βρετανική εκδοχή της αγγλικής θα είναι μια όλο και πιο σπανίως χρησιμοποιούμενη διάλεκτος το αισιόδοξο σενάριο τώρα. Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, εμεί οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ολλανδοί, οι Πολωνοί και ούτω καθεξή έχουμε κάνει προσπάθειε και βάλαμε και τα παιδιά μα να μάθουν καλά δύο άλλε γλώσσε τουλάχιστον επιπλέον τη μητρική του γλώσσα και ίσω να καταλαβαίνουν και κάτι από κάποιε άλλε γλώσσε. Οι μόνε εξαιρέσει είναι, είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι συνήθισαν να μιλούν όλοι οι άλλοι τη γλώσσα του λίγο πολύ καλά και έτσι σταματήσαν εδώ και καιρό να μιλούν ξένες γλώσσες. Καθώς όμως είναι και λογικοί άνθρωποι, κάποια στιγμή θα αντιληφθούν ότι με αυτόν τον τρόπο και η σκέψη του και η αντίληψή του στενεύουν και ότι η έμμονη μονογλωσία τους σημαίνει ταυτόχρονα και πολύ περιορισμένη θεώρηση σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκος και καθώ δεν θέλουν να παραμένουν σε περιορισμένα όρια θα ε, στραφούν πολύ γρήγορα και εντατικά στην εκμάθηση τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών και θα φροντίσουν και τα παιδιά του να μαθαίνουν τι ε, άλλε δύο γλώσσε. και έτσι όλοι στην Ευρώπη από, τα 50, από 50 100 ετών θα μπορέσουν να έχουν μια ποικιλία πολιτιστική, γλωσσική έναν πλούτο και μια δημιουργικότητα. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτό που μετράει σοβαρά δεν μπορεί να καταμετρηθεί και αυτό που μπορεί να καταμετρηθεί δεν μετράει πάντα απαραίτητα. Νομίζω ότι ήταν λόγια του Αϊνστάιν. Έχουμε λοιπόν πολλούς καλούς λόγους να συνεχίσουμε να προάγουμε την πολυγλωσία και την ευρυγλωσία στην Ευρώπη, άλλοι λόγοι οικονομικοί, άλλοι προ το συμφέρον μια πιο ισχυρή δημοκρατία. Ενώ άλλοι είναι μη προσμετρήσιμοι. Ο, Βρετα... ο Ιρλανδό ποιητή Σαμοσίνη, που έχει βρεβευτεί με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνία του 1995, μετρική γλώσσα την αγγλική και που απεβίωσε πέρυσι, είχε μιλήσει για τη σημασία που θεωρούσε πω έχει ε, για τον ίδιο ναι, η εκμάθηση της Ιρλανδικής, μιας γλώσσας που δεν έχει ε, οικονομική αξία έξω από την Ιρλανδία. Με ιδέες που είναι αντίστοιχε με αυτές του Λομπιάνκο αλλά σε μια γλώσσα πολύ πιο ποιητική μας λέει με επιχειρήματα που ε, αφήνουν κατά μέρο την ομοιογενοποίηση και λέω τα λόγια του όπως, τα, όπως μας τα άφησε, το να μην μάθει κανείς την Ιρλανδική σημαίνει να χάνει την ευκαιρία να καταλάβει πώς ήταν αυτή η χώρα και τι σημαίνει αυτή η χώρα, αλλά και τι, τι καλύτερο μέλλον μπορεί να φέρει σε αυτή η χώρα. Σημαίνει να κόψει τις ρίζες του, σημαίνει να χάσει την αυτοαντίληψή του, την άλληλο αντίληψή του, την ε, πνευματική του και φαντασιακή του ανάπτυξη, την πολιτιστική του διαφορά, την πολιτική του ανεκτικότητα. Σα ευχαριστούμε πολύ καθηγήτρια Γκάλαχερ και ελπίζουμε ότι το αισιόδοξο σενάριο του καθηγητού Στίκλ θα είναι αυτό το οποίο θα επιβληθεί στα επόμενα χρόνια. Με την αισιόδοξη πρόπτικη λοιπόν για όλους μας είμαι βεβαία ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για την καθηγήτρια Κάλαχερ αλλά ίσως να χρειαστεί να καθυστερήσουμε τις ερωτήσεις αυτές και να τις αφήσουμε για το μεσημεριανό. Έχουμε εδώ την πρώην Γενική Αρμόδια Επικεφαλής των Διερμηνέων του State Department των Ηνωμένων Εθνών. Έχει συνεργαστεί στην ανάπτυξη του τμήματος διερμηνίας στο Πανεπιστήμιο του Maryland. Είναι από τους ε, προτεργάτες της πρωτοβουλίας HINTS, Επικεφαλής ε, Υπηρεσιών Διερμηνίας των Διεθνών Οργανισμών. Σας καλωσορίζουμε εδώ και παρακαλώ να μας πείτε εσείς τι αποκομίζετε από τη σημερινή συνεδρίαση, τι συμπεράσματα μπορείτε να διατυπώσετε, παρακαλώ. Προσοχή. start... Θα μιλήσω αγγλικά τώρα και θα ξεκινήσω με κάποιες λέξεις που τρομοκρατούν κάθε διερμηνέα. Θα σας πω ένα αστείο. Αυτή είναι η εισαγωγή που τρομάζει κάθε διερμηνέα. Κάποιος και πρώτη φορά φυλακίζεται. Είναι κλεισμένο στο κελί του και κλείνουν τα φώτα στο κελί. Πηγαίνει λοιπόν προς τα κάγκελα και κραυγάζει. Δώδεκα. Αρχίζουν και απαντούν με σπασμωδικά γέλια όλοι οι υπόλοιποι τρόφιμοι της φυλακής. Κάποιος άλλος φωνάζει. Τέσσερα. Και πάλι ξεκαρδίζονται στα γέλια όλοι οι έγκλειστοι στη φυλακή. Μπερδεύτηκε ο φυλακισμένος, γυρίζει προς τον α, συγκάτοικο του στο κελί και το ρωτάει «Συγγνώμη, μπορείς να μου εξηγήσει τι συμβαίνει» Εκείνος του λέει Μερικοί είμαστε πολύ καιρό στη φυλακή, οπότε έχουμε ένα ολόκληρο ρεπερτόριο αστείων. Τα έχουμε επαναλάβει τόσες φορές, απλώς τα νούμερα αναφέρουμε και γελάμε. Οπότε ξανασπέβδει στα κάγκελα και ε, φωνάζει. 17 ησυχία, νεκρική σιγή. Γυρίζει λοιπόν στο, στον συγκάτοικό του και του λέει τι γίνεται, το αστείο υπαριθμό 17 δεν ήταν καλό. Όχι καλό ήταν, του λέει ο άλλος. Αλλά δεν έχουν όλη την ικανότητα να δίγονται ανέκδοτα. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία. Θέλω να ευχαριστήσω την Όλγα Κοσμίδου για την ε, πολύ καλή ε, πρωτοβουλία που ανέλαβε, που ήταν μία ακόμη σε μία σειρά αξιόλογων πρωτοβουλειών που έχει λάβει. Και σας παραπέμπω στο πρόγραμμα που λάβαμε. Παγκόσμιο Φόρουμ Διερμηνίας. Wow! και επιτυχία της αριστείας και της αρτιότητας στη διερμηνία των συνεδριάσεων. Διπλό wow. Και ακούσαμε καταπληκτικούς ομιλητές το τελευταίο διήμερο. Ο καθηγητής Βάιμπελ μας μίλησε για την αυτόματη, τη μηχανική διερμηνία. Άρχισα να τρέμω στην καρέκλα μου, δεν ξέρω εσείς πώς αισθανθήκατε. Αλλά πολύ γρήγορα μας εξήγησε ότι σε καμία περίπτωση θέλουν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη προσπάθεια, απλώς να βοηθήσουν, να στηρίξουν την επικοινωνία. Και χαίρομαι που χρησιμοποίησε τον όρο επικοινωνία. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η πεμπτουσία της διερμηνίας. Η διερμηνία δεν αφορά τις γλώσσες. Δεν μιλούμε εδώ για μετάφραση και διερμηνία σε τελική ανάλυση. Μιλούμε πάνω απ' όλα για επικοινωνία. Και επιμένω σε αυτό. Ξέρω βέβαια ότι όλοι πεινάτε και θέλετε να σπεύσετε να φάτε. Γι' αυτό και τονίζω ότι δεν μιλάμε εδώ μόνο για γλώσσες και λόγο και ομιλίες, αλλά για επικοινωνία. Μας μίλησε επίσης για αριστεία, για την πρόκληση της στοχευμένης εξάσκησης, της επισταμένης εξάσκησης. Και φυσικά μόνο ο Θεός ξέρει τι προσπάθεια κάνουμε. Είχα, ανακάλυψα δύο κουτιά με γλωσσάρια από το 75 τα κρατούσα από τότε. Αλλά σκέφτηκα, ο κόσμος έχει αλλάξει, τεχνολογίες, δεν κρατάμε πια γλωσσάρια σε χαρτί. Ο κύριος ε, Καλβέ, ο κύριος μίλησε για την ε, ε, γλωσσική πλευρά της παγκοσμιοποίησης και μας αποκάλυψε τη βαρομετρική πίεση που ισχύει στην προσπάθεια ταξινόμησης των γλωσσών. Και το είδαμε και αυτό και στη συζήτηση που ακολούθησε. Και αισθάνομαι μια σπάνια χαρά και απόλαυση όταν ακούω τη, τις ομιλίες του κυρίου του καθηγητού Άντελμαν που μίλησε για την ευρωβιολογία στη Διερμηνία. Και μας είπε ότι έχουμε και ερπετοειδή εγκέφαλο που είναι πολύ αθαρρυντικό γιατί εγώ το ήξερα ότι έχω τέτοιο. Επίσης, η κυρία, οι δύο ερευνήτρες μας μίλησαν για, την, το σχετισμό μουσικών και διερμηνέων και ότι <laughs> μας είπαν ότι οι διερμηνείς έχουν πανκ εγκέφαλο. Ακούσαμε και για την ανάγκη της πολυδιεργασίας, του multitasking. Μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσες α, ταυτόχρονες ενέργειες επιτελούμε και μάλιστα περιμένουμε από εμά να τα κάνουμε όλες με άρτιο τρόπο. Λέω στους διερμηνείς ότι μπορεί να είναι κανείς ο καλύτερος διερμηνέας του κόσμου, πολύπυρος, αλλά και μία φορά να αποτύχει, κάηκε. Το μέλλον του σφραγίστηκε. Αυτό που αποκόμισα από κάτι που είπε η συνάδελφος Λουαζό, είναι ότι είναι σημαντικό να έχουμε το σκοπό μας κατά νου. Δηλαδή ότι δεν είμαστε ένα απλό άθροισμα των συνιστοσών. Είμαστε όλοι συνιστώσει μαζί, αλλά και ταυτόχρονα ο σκοπός μας. Και ποιο είναι ο σκοπός μας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας. Η δόκτωρ Ολιβέρα μίλησε για την προσαρμοστικότητα και πώ θα την επιτύχουμε. Βέβαια, αυτό είναι σημαντικό. Πώς θα επιτύχουμε την προσαρμοστικότητα. Η καθηγήτης Γκάλαχερ μίλησε για την ε, πολυγλωσία σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, τη lingua franca, τη μονογλωσία, τη μονογλωσσικότητα και σε μία από τις παραθέσεις που έκανε, σε ένα από τα αποσπάσματα, ήταν πολλά τα ενδιαφέροντα, σε ένα είπε είναι σημαντικό να διαβάζει κανείς πίεση ε, σε μία γλωσσική ζώνη. Ποιήση, και λογοτεχνία. Και μία και μόνο γλώσσα μας είπε δεν αρκεί για να ικανοποιηθούν οι γλωσσικές και κυρίως οι επικοινωνιακές μας ανάγκες. Θα ήθελα να επανέλθω λοιπόν στο πρώτο ζητούμενο και στο πρώτο σχόλιο που άκουσα χθες η Όλγα Κοσμίδου μας μίλησε για το θαύμα της διερμηνίας. Καθόμαστε εδώ, συνεδριάζουμε εδώ και είναι τόσο μεγάλη απόλαυση, χαρά αλλά και τιμή που συγκεντρωνόμαστε όλοι σε μία και μόνο αίθουσα. Τι ωραία που θα ήταν να είχε συμβεί αυτό πριν από 30-35 χρόνια αλλά πραγματικά τότε θα ήταν ε, πολύ πρωτόγνωρο και πρωτοφανές και πραγματικά κοιτάω γύρω μου και αγαλιάζω. Η ταυτόχρονη διερμηνία ξεκίνησε τον 20ο αιώνα, το γνωρίζουμε. Και τώρα αναλύουμε το φαινόμενο λεπτομεριακά, κάνουμε μία τομή και προσπαθούμε να δούμε ε, πώς ε, λειτουργεί. Αλλά δεν δεν ξέρουμε πραγματικά. Όπως είπε και κάποιος στο Shakespeare in Love στην ταινία, δεν ξέρουμε. Είναι ένα θαύμα. Και στην διερμηνία, για να επιτύχουμε την αριστεία και την αρτιότητα, δεν είναι να μάθουμε μια τριπλή περιστροφή, ένα σάλκο ή να μάθουμε γοεδελικά. Είναι ενίσχυση της μνήμης μας. Δεν είναι σαν να μαθαίνουμε σκάκι και να απομνημονεύουμε μια ακολουθία κινήσεων. Αυτό το κάνουν και οι υπολογιστέ. Υπάρχει και μια άλλη δυσκολία για την εξασφάλιση της αριστεία στη Δερμηνία. Το επισήμαναν και ο κύριος Ερβέντελμαν και ο καθηγητής Έριξον. Ποιο μπορεί να αξιολογήσει, ποιο μπορεί να καταμετρήσει την απόδοση του Διερμηνία. Σίγουρα όχι το ακροατήριο. Σίγουρα όχι ο πελάτης. Μερικές φορές ε, οι πελάτες ε, συμπαθούν τους διερμηνείς γιατί μπορούν να δουλεύουν 12 ώρες συνέχεια ή να οδηγήσουν ή να καθαρίζουν τα παράθυρα. Γελάτε, γελάτε, αλλά και αυτό συμβαίνει. Και είναι πραγματικά λυπηρό. Μερικές φορές δυστυχώς οι μόνοι που μπορούν να αξιολογήσουν ένα διερμηνέα είναι οι ίδιοι διερμηνείς. Αυτό σημαίνει το να εμπλέκονται οι διερμηνεί στη διαχείριση της διαρμηνίας. Και εγώ είμαι κάποιος ο οποίος είχα εμπλακεί σε μια οργάνωση όπου οι διερμηνείς διαχειριζόντουσαν τους διερμηνείς. Και οι υπόλοιποι έπρεπε να χρειαστεί να μάθουν γρήγορα τι ήταν η διερμηνία. Και αυτό συμβαίνει και για μας. Οι καλύτεροι φίλοι που είχαμε ποτέ ήταν ε, οι υψηλά κυβερνητικοί ιστάμενοι οι οποίοι κατανοούσαν πόσο καλά οι διευμηνείς ετοιμάζουν τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν. Θα επαναλάβει κάτι το οποίο είπε ο Will και σε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Έριξον. Ο κ. Ντουρόν είπε ότι εμείς είμαστε αυτό το οποίο επανειλημμένα κάνουμε. Η αριστεία δεν είναι μία απλή πράξη, αλλά είναι ένα συνήθιο. Και σαν διερμηνής η αριστεία, η βέλτιστη πρακτική πρέπει να γίνει συνήθιο. Γιατί εμείς επικοινωνούμε. Γιατί όπως είπε και η Δόκτωρα Λιβέιρα και η κυρία Λουαζό, εμείς στην ουσία γράφουμε ωραία μουσική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας προκαλέσω να κάνετε έναν κατάλογο το τι πρέπει να κάνει κανείς ε, σαν διευμηνέα. Σας περάσουμε στην πολλαπλή δραστηριότητα, ε, στην διεργασία. Τι πρέπει να κάνει ο διευμηνής, τι θα χρειαστεί να κάνει ο διευμηνέας στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Το να επικοινωνεί κανείς είναι κάτι το καινούριο και κάτι το παλιό μαζί, όπως και η διευμηνία και οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η νέα γενιά είναι τεράστιες. Ο κόσμος είναι πολύ μικρότερος από ό,τι ήταν ποτέ και θα γίνει ακόμα πιο μικρός. Οι νέες γλώσσες. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πριν 20 χρόνια ότι θα μιλάμε μέσω του texting, με hashtags. Δεν τα καταλαβαίνω, ακόμα και σήμερα. Θα σας δώσω ένα μικρό κατάλογο και θα πρέπει να το σκεφτείτε. Γιατί εσείς είσαστε το μέλλον της διευμηνίας και αυτό το οποίο εσείς θα κάνετε θα καθορίσει το αν θα βουλιάξουμε ή θα επιβιώσουμε. Προσοχή. Φυσικά ο διευμηνέας δεν ακούει μόνο λέξεις, στην ουσία η οικοδομή της λέξης που ακούει. Μια μηχανή δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει, δυσκολεύομαι να το πιστέψω διέστηση. Είναι ένα μέσο η γλώσσα στα πλαίσια της επικοινωνίας. Είναι ακριβώς ε, το σημείο εκκίνησης. Πώς να επικοινωνήσει κανείς σηκώνοντα το βλέφαρό του σαν παράδειγμα. Η σιωπή πώς να την διερμηνεύσει. Η διακριτικότητα επίσης. Ξέρει κανείς οπότε έφτασε η στιγμή του να δείξει τάκτ και εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό όργανο Πολλή διερμηνία γίνεται σε πολιτικό επίπεδο βέβαια. Πρέπει να είναι αόρατος ο διερμηνέας. Να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχει για να φωτίζει ε, και να τονίζει αυτό το οποίο λέει ο, ο μιλητής. Οι διερμηνείς είναι ηθοποιοί οι οποίοι δεν έχουν μια σκηνή στη διάθεσή τους και στο τέλος δεν τους χειροκροτεί κανείς. Είναι μια μάλλον αχάριστη δραστηριότητα το να είσαι διαμηνέας. Πρέπει να είναι ακέραιοι, πρέπει να είναι όπως είπαμε διακριτική. Πρέπει να αποφεύγουν το να βάζουν και το δικό τους. Πρέπει να ελέγχουν τις γλώσσες τους όπως είπε και η Αν Αυτό ξεκινάει με τη μητρική σας γλώσσα και πάρα πολλοί φοιτητέ το ξεχνάνε. Το θέμα δεν είναι να μαθαίνουν γλωσσάρια και καταλόγους λέξεων. Αν δεν μπορεί να μιλήσει κανείς καλά στη μητρική του δεν έχει κανένα νόημα να είναι σε καμπίνα διαρμηνίας. Να έχει τη δυνατότητα να ομιλεί σε δημόσιο. Δεν αρκεί κανείς ε, να είναι ικανός να μεταφράζει έναν καλό ομιλητή, αλλά πρέπει να μεταφράζει και τον κακό μιλητή. Δεν θα ήθελα να ακούω ένα κακό μιλητή για μισή ώρα. Αυτό έχει σχέση και με την εκπαίδευση φωνής και για τις ασκήσεις για την διαδοχική που είναι δύο διαφορετικές ικανότητες και στον τρόπο έκφρασης και όπως είπε ένας από τους συναδέλφους χθε και το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους, πάρα πολλούς, πρέπει να παίζει κανείς το ρόλο του, πρέπει να κάνει θέατρο, να υποδίεται γιατί η δουλειά του διερμηνέα είναι πολύ κοντά σε αυτά που έλεγε ο Στανισλάβσκι όταν έλεγε ότι έχει ανάγκη ο ηθοποιός να βρει τον στόχο. Οι διερμηνείς δεν αναζητούν καν τον συγκεκριμένο στόχο. Πολιτισμός, εκπαίδευση, ενημέρωση, να γνωρίζουν τα διάφορα επίπεδα της, ε, ε, του μηνύματος που θέλει ο μιλητής να μεταφέρει. Και επαναλαμβάνω, Όλα έχουν σχέση με την επικοινωνία. Για να στραφούμε λοιπόν προς το μέλλον θα πρέπει να δούμε την ε, δεξιότητα, την υπεροχή σε αυτή, την αριστεία σε αυτό το επάγγελμα που τόσο αγαπάμε. Τι ψάχνουμε εδώ λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η σημασία του αυτού που έχουμε εδώ, αυτή της ένωσης οργανώσεων διεθνών, εθνικών, διεθνικών, διοεθνικών, πανεπιστημίων που κάνουν τόσο καταπληκτική δουλειά. Μια ομαδική δουλειά, μια ομαδική δραστηριότητα, όπως είναι και η διερμηνία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οι διερμηνείς δεν είναι μηχανές. Είναι σημαντικές οι συνθήκες εργασίας μην επιτρέψετε να υπονομευθούν από οποιαδήποτε γραφειοκρατική επιλογή ή διερμηνείς, μην επιτρέψετε τη διερμηνία να πέσει ποτέ στο ρόλο του πιο αδύναμου κρίκου. Κάποιος θες μου έλεγε μια ιστορία, ότι να ένας διερμηνέας φτάνει στην καμπίνα για με τέσσερις γλώσσες. Όπως προχωράμε θα πρέπει να θυμόμαστε και κάτι άλλο που έχουμε κοινό για το επέγγελμά μας. Το πάθος. Και ελπίζω να μπορώ να σας το μεταδώσω. Μας νοιάζει η διερμηνία, μας νοιάζει το μέλλον της, μας νοιάζουν οι νέοι αυτοί οι οποίοι πονούν και καταπονούνται για αυτήν. Το είδαμε άλλωστε απτά αυτές τις δύο μέρες, διότι η ποιότητα και η αριστεία της διερμηνίας θα προσδιορίσει και το μέλλον της και άρα εξαρτώμεθα από όλους εσάς. Τα μόνα λόγια που έχω να σας απευθύνω είναι ας φύγουμε από αυτό το υπέροχο κέντρο συζητήσεων και να πάμε να βγούμε και να κάνουμε μια υπέροχη μουσική όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το μόνο μπορώ να συμπληρώσω είναι ένα διπλό wow. Δεν υπέροχα αυτά που μας είπες και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας όλων σε αυτές τις δύο ημέρες των εργασιών. Πριν προχωρήσουμε όμως περισσότερο για τα τελευταία θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Όλγα Κουσμίδου, Γενική Διευθύντρια. Θα πω εγώ τα εξής όμως πρώτα. Έχουμε ένα ε, γεύμα σε μπουφέ εδώ έξω από την αίθουσα. Για το απόγευμα έχουμε προβλέψει δύο workshops για τους course leaders στην αίθουσα 6Q1, στον ίδιο όροφο προς τα αριστερά όπως θα βγείτε. Το πρώτο έχει να κάνει με, τα, με τις υποτροφίες, τις ε, ενισχύσεις, τις πανεπιστημιακές και ενημέρωση για αυτές, αλλά θα δώσουμε και τη δυνατότητα για διμερείς επαφές, ερωτήσεις σχετικές ε, με τις σχετικές ενισχύσεις. Και το δεύτερο ε, workshop έχει να κάνει με τις εξαποστάσεως, με την στη διδασκαλία υπό την Κατερίνα Δάρα πάλι στην ίδια αίθουσα, θα αρχίσει λίγο αργότερα. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για την παναφρικανική διάσκεψη διερμηνίας και μετάφρασης θα ξεκινήσει η συνεδρίασή της στις 2.45 εδώ στην αίθουσα που βρισκόμαστε, 6Q2. Η Πάτση όμως μίλησε πολύ για το πάθος η Όλγα νομίζω έχει πάρα πολύ πάθος για το επάγγελμα αυτό και θα μας μιλήσει τώρα για το Οικουμενικό Δίκτυο Αριστείας για το Μέλλον. Όλγα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Σουζάν. Μετά την παρέμβαση κατηγορίας διπλού wow της Πάτσι, λίγα μου μένουν εμένα να πω, να πω νομίζω. Θέλω απλώς να της πω ότι συμμερίζομαι το πάθος της. Το πάθος της για αυτό το επάγγελμα Τόσο μάλιστα που όταν κάποιος που δεν με πολύ γνωρίζει με ρωτάει τι δουλειά κάνω και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια που δεν έχω μπει σε καμπίνα, η απάντηση που δίνω πάντα είναι διερμηνέας. Και για μένα αυτό αποτελεί τίτλο τιμής. Είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό επάγγελμα. Σας βάζει σε ένα, άλλο κόσμο. Πολύ συχνά δεν λέω όταν συναντώ νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια και στους οποίους θέλω να αφυπνίσω και να μεταλαμπαδεύσω αυτό το πάθος τους λέω λοιπόν ότι το επάγγελμα αυτό σε υποχρεώνει να αναλύσεις το μήνυμα για να μπορέσει να το μεταδώσεις. Το επάγγελμα αυτό, τους λέω, σε υποχρεώνει να μπει μέσα στο μυαλό του ομιλητή. Και με αυτόν τον τρόπο το επάγγελμα αυτό σε βοηθάει να ξεχωρίζεις το γνήσιο, το αυθεντικό από το κάλπικο. Και προσοχή στο μέλλον ποιον θα παντρευτείτε. Κι όμως το επάγγελμα αυτό δεν έχει επαρκή αναγνώριση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν πολλά άλλα επαγγέλματα όπου ο καθένας να μπορεί να ισχυριστεί πως είναι διερμηνέας ή μεταφραστής. Δικηγόρος πάντως δεν μπορεί να το κάνει. Και ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι γιατρός. Ναι. Αλλά ο καθής μπορεί να πει είμαι μεταφραστή ή είμαι διερμηνέας. Με πολύ κακά, πολύ κακές επιπτώσεις για το επάγγελμα εν τέλει. Αρκεί, όπως το είπε και η Πάτση, και ισχύει και για τον αληθινό διερμηνέα, για τον γνήσιο διερμηνέα. Μία φορά να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η διερμονία δεν θεωρείται απόλυτο ικανοποιητική, για να καταλήξουν οι στο συμπέρασμα ότι τελικά δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το επάγγελμα και τόσο απαραίτητο. Και εγώ ύστερα από τόσα χρόνια στο επάγγελμα διαρκώς καταπλήσωμαι όταν βλέπω ότι αυτοί που ετοιμάζουν μια μεγάλη διάσκεψη μπορεί να σκεφτούν τα πάντα, την αίθουσα, τους τεχνικούς, την τεχνολογία, την αναψυχή, ε, την εστίαση, και μετά θα πάει το μυαλό του στη διερμηνία. Τελευταία στιγμή τι θυμούνται. Και όπως εν γέννη έχουν ήδη μπει σε μεγάλα έξοδα, προσπαθούν να κάνουν οικονομία από τη Διερμηνία. Ενώ δεν ζητούν ε, από, τον, από το catering ε, να δώσει μπαγιάτικο κρέας για να γίνει πιο οικονομικό το φαγητό ζητούν στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες διερμηνίας αντί για έξι διερμηνίες που θα απαιτούνται να δώσει μόνο τέσσερες ή αντί για επτά ώρες να δουλέψουν εννιά ώρες οι διερμηνίες. Με απασχολεί λοιπόν το γιατί. Οφείλεται άραγε αυτό στο ότι όπως μας λένε τα αγγλικά είναι πλέον τόσο διαδεδομένη γλώσσα που η διερμηνία δεν είναι πλέον απαραίτητη. Μήπως η διερμηνία σιγά σιγά γίνεται κάτι το οποίο βρίσκεται γιατί το έχουμε συνηθίσει, γιατί κάπως μας βολεύει. Καλού κακού. Όχι. Η καθηγήτρια Γκάλαχερ μας είπε ότι είναι λιγότεροι από 50% οι Ευρωπαίοι εκείνοι οι οποίοι καταλαβαίνουν σε καλό επίπεδο τα Αγγλικά. Και μάλιστα σε ορισμένες χώρες της Ένωσης. Ούτε το 20% του πληθυσμού δεν καταλαβαίνει καλά τα Αγγλικά. Θέλουμε λοιπόν να αποκλείσουμε όλους αυτούς τους πολίτες επιβάλλοντας μία κοινή γλώσσα. Και μαζί με αυτήν και μία ενιαία γλώσσα. Ε, μία ενιαία σκέψη. Μήπως την ώρα που όλοι διερωτώνται γιατί ο πολίτης έχει τις αποστάσεις του από την πολιτική, γιατί πια δεν πάει να ψηφίσει ο πολίτης. Θέλουμε πράγματι να τον αποκλείσουμε τον πολίτη σε τέτοιο βαθμό. Θέλουμε πράγματι τα συνθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενωμένη στην ε, ποικιλία, στην πολυμορφία να γίνουν ε, γράμμα κενό. Και όταν λέμε όλοι μιλάνε αγγλικά. Πρώτη γλώσσα τα αγγλικά. Μα ξεχνάμε να πούμε ακόμα και εδώ μέσα ότι τα αγγλικά είναι η πρώτη ξένη γλώσσα. και δεν είναι, οπωσδήποτε δεν είναι η πρώτη γλώσσα, μητρική γλώσσα στον πλανήτη. Μπορεί να είναι η πρώτη σε χρήση ως μητρική γλώσσα. Μου λένε μην προσπαθήσει να ανατρέψει το ρεύμα. Ναι, η ιστορία όμως μας διδάσκει ότι υπήρξαν πολλές κοινέ γλώσσες, πολλές Λίγκου φράγκε, τα ελληνικά, τα ραμαϊκά, τα λατινικά, τα γαλλικά. Τώρα τα αγγλικά. Και ποιος μπορεί μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος διαρκώς κινείται και που παρουσιάζεται τις μεταλλάξεις θα μπορούσε να προβλέψει τη μορφή που θα έχει ο προσοχής αιώνας και ποιες θα είναι οι κοινέ γλώσσες, η lingua franca. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι μετά την βιομηχανική επανάσταση και επανάσταση των επιστημών θα σημειωνόταν επάνωδος στην θρησκεία. Πρέπει πραγματικά να μάθουμε ότι αυτό το οικουμενικό χωριό δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αποκλείοντας ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών του. Και τη στιγμή όπου τα κινήματα των πολιτών, μετακινήσεις των πολιτών καλύτερα, για λόγους όχι απλώς τουρισμού, αλλά μετακινήσεις για λόγους ανθρωπιστικής κρίσεως, πλημμυρών, φυσικών καταστροφών και άλλους. Σημαίνουν ότι δεν υπάρχει πλέον χώρα με καθαρό φιλετικό χαρακτήρα ή χώρα στην οποία ομιλείται μόνο μία γλώσσα από όλους τους πολίτες της. Μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε τα γλωσσικά επαγγέλματα που είναι η μόνη εγγύηση μιας δημοκρατικής αντιμετώπισης αυτών των πολιτών. Μπορούμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα στον υπήκο μιας άλλης χώρας να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα χωρίς να του προσφέρουμε και τη δυνατότητα να περάσει από δικαστήριο εάν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη να περάσει την ακροματική ε, διαδικασία στη δική του γλώσσα ή να πάει να τον κοιτάξουν σε ένα νοσοκομείο εάν δεν μπορεί να εξηγήσει τα συμπτώματα που αισθάνεται στη δική του γλώσσα. Ναι βεβαίως και αυτό συνεπιφέρει κόστος. Αλλά αυτό είναι το κόστος της δημοκρατίας, έτσι λέγεται. ή για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από μερικά χρόνια, όταν ένας δημοσιογράφος του είπε «Ω, η μετάφραση, η διερμηνία κοστίζει τόσο πολύ. Πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε οικονομίες από αυτούς τους πόρους». Ε, μα του απάντησε αυτός ο αντιπρόεδρος Επιτροπής «Και οι εκλογές κοστίζουν. Τι έχετε να μου πείτε». πρέπει οι γλώσσες να μπουν στο ίδιο το επίκεντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν ρωτήσετε τους οικονομικούς φορείς ποια είναι η πιο σημαντική για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις οικονομικές συναλλαγές γλώσσα, ποια είναι η μία πιο σημαντική για τις οικονομικές συναλλαγές γλώσσα, είναι η γλώσσα του αγοραστή. Δεν είναι μια οικουμενική γλώσσα. Και αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι έμποροι. Στη χώρα μου. Όλες οι πινακίδες των καταστημάτων δεν, γράφονται, δεν αναγράφονται πια στα αγγλικά, αλλά στα ρωσικά, λόγω του τουρισμού. Εδώ και χρόνια. Και να μην σας μιλήσω για την Κύπρο, όπου σχεδόν τα πάντα αναγράφονται στα ρωσικά. Και σιγά αρχίζουμε, σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε και κινέζικα. Υπάρχουν λοιπόν τα γλωσσικά επαγγέλματα που και η παρουσίαση του κυρίου, του δόκτωρα Βάιμπελ με καθησυχάζει ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να έχουν το μέλλον τους τα, τα γλωσσικά επαγγέλματα και θα πρέπει ο καθένας να βρει τη θέση του θα πρέπει να εξασφαλίσουμε για το κάθε επάγγελμα να το περιγράφουμε σωστά γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει συνήθως ποια είναι η διαφορά μεταξύ μετάφρασης και διερμηνίας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διερμηνίας επαφής και διερμηνίας συνεδρίων, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τον κόπο, να εξηγήσουμε. Και όπως είπε και η Πάτση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι η διερμηνία παρεμπιπτόντως μόνο έχει σχέση με τις γλώσσες. Οι διερμηνείς δεν είναι λεξικά με πόδια. Πολύ συχνά μου λένε «Α, αυτό πώς το λες στα ελληνικά, πώς το λες στα ισπανικά». Ιδέα δεν έχω. Την ώρα που μεταφράζω ως διερμηνέα στην καμπίνα, βρίσκω τον τρόπο να το μεταφέρω. Αλλά χωρίς συμφραζόμενα, αν με ρωτήσετε πώς ε, τη λες αυτή τη λέξη, πώς λες την άλλη λέξη, δεν μου έρχεται. Και κάποιος που δεν είναι του επαγγέλματος, διερωτάται, μα τι διερμηνέας να είναι αυτή, άμα δεν μπορεί να μου πει μια λέξη. Έλεγα λοιπόν ότι έχει μέλλον και είμαι πεπισμένη πως έχει μέλλον Για να είναι λαμπρό λοιπόν το μέλλον αυτό, χρειαζόμαστε τη δική σας συνδρομή. Γι' αυτό και η ιδέα του Οικουμενικού Φόρουμ. Διεθνείς οργανισμοί. Οι διεθνείς οργανισμοί τη δουλειά τους δεν μπορούν να την κάνουν χωρίς τη δική σας συνδρομή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν δεν σας εξηγήσουμε πως το επαγγελματικό επίπεδο που ζητάμε δεν αντιστοιχεί πάντα στο επίπεδο των πανεπιστημιακών επιδόσεων που απαιτούνται για να πάρει κανείς ένα δίπλωμα. Άρα, μια διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγές μεταξύ ημών και ημών, έτσι ώστε και εμείς να αντιληφθούμε καλύτερα τα δικά σας προβλήματα και εσείς να αντιληφθείτε καλύτερα τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες είναι απαραίτητη. Ιδάλλως, σε ένα επάγγελμα με μέλλον κινδυνεύεται να καταρτήσετε ανέργους στο μέλλον. Και αυτό θα ήταν κρίμα γιατί και εμείς θα μείνουμε χωρίς διερμηνείς και εσείς θα καταρτίζετε διερμηνείς που δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Γι' αυτό και είχαμε αυτήν την ιδέα για το φόρουμ. Και σε ορισμένα πανεπιστήμια, εδώ και καιρό, έχουμε διαπιστώσει πως μηχανικοί επικοινωνούν με, την, ε, με τη βιομηχανία, με το χώρο της παραγωγής. Κάνουν την εκπαίδευση τους στην πρακτική εκεί και τους δίνει η βιομηχανία το μέτρο του επίπεδου επιδόσεων που χρειάζεται. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις αξίες. Το επίπεδο. Υπογραμμίζουμε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται προφανή, αλλά που είναι τόσο μα τόσο απαραίτητα. Η Πέρση μίλησε για την ε, μητρική γλώσσα, τη γλώσσα προς την οποία ε, εκφράζεται ή στην οποία εκφράζεται ο διερμηνέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας τα πανεπιστήμια, να εξηγείτε και να λέτε στους φοιτητές σας πως υπάρχει δεοντολογία, πως δεν μπορούμε να μεταφράζουμε προς οποιαδήποτε γλώσσα. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τη διερμηνία είναι το περιτύλιγμα της σκέψης μας. Το περιτύλιγμα της σκέψης. Και πρέπει αυτό το περιτύλιγμα να είναι διαμορφωμένο ανάλογα με τη σκέψη και όχι η σκέψη να προσαρμοστεί στο περιτύλιγμα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο διερμηνέας ο οποίος εργάζεται προς μια γλώσσα που δεν κατέχει πραγματικά, δεν μπορεί να εκφράσει το προϊόν και δίνει μόνο αυτό που του επιτρέπει να προσφέρει το περιτύλιγμα. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το φόρουμ αυτό το βλέπω ως μόνη δυνατότητα να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε το επάγγελμα. Θα έχετε ασφαλώς παρατηρήσει ότι αντίθετα με όσα συνέβαιναν στο παρελθόν υπήρξε διάλογος μεταξύ αυτών που έκαναν τις παρουσιάσεις τους διεθνούς επίπεδου ε, ειδικού μας επιρογνώμονες, τους οποίους και ευχαριστώ που απεδέχθησαν την πρόσκληση και ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν και βρίσκονται ακόμη εδώ, που όμως δέχθηκαν και τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Γιατί μόνο χάρη σε αυτό το διάλογο μπορούμε να συνεχίσουμε. Πριν από 20 περίπου χρόνια, ο Νοέλ Μόιλε, τον οποίο και ευχαριστώ, η Νοέλ Μόιλε που και ευχαριστώ που βρίσκεται εδώ, με πήρε κατά μέρο και μου ψήφισε την ιδέα να δημιουργηθεί το, ένα ευρωπαϊκό Masters για την διερμηνία συνεδριών. European Masters on Conference Interpretations με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δέχθηκα, εξεργαστήκαμε περισσότερο την ιδέα, την ξεκινήσαμε. Το βρέφος αυτό προχώρησε τόσο καλά που πια δεν έχει ανάγκη νονές και νονούς. Είχε τεράστια επιτυχία. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος λογότυπος. Αλλά είχε ως όρια τα σύνορα της Ευρώπης. Κρίμα διότι ζούμε όλοι σε ένα οικουμενικό χωριό, σε ένα παγκόσμιο χωριό. Δεν μπορεί πια κανείς να λέει ότι μπορεί να αρκεστεί στις 24 γλώσσες της Ευρώπης. Έστω και αν αυτές θεωρούνται υπερβολικά πολλές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνθήκη της Λισαβόνας μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή σε κύριο συνομιλητή στη διεθνή σκηνή. Αναπτύσσει εταιρικέ σχέσεις και με άλλα, με άλλες κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, όπως τον χωρό Νακέ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τη Euromed, όπου τα αραβικά, τα εβραϊκά, τα τουρκικά είναι πολύ σημαντικές γλώσσες. Τελευταία φτάνει, καταφτάνει και η Euronest. Με τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα σημαντική τη ρωσική γλώσσα. Έχουμε όλο και περισσότερη ανάγκη τις γλώσσες αυτές γλώσσες οι οποίες ήταν ε, περιορισμένες σε χρήση μόνο στην οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους φίλους από τα Ηνωμένα Έθνη που είναι παρόντες εδώ και οι οποίοι μας βλέπουν. ως συνεταίρους και συνεργάτες και όχι ως ανταγωνιστές. Όντως αναζητούμε την αριστεία. Και εκείνοι και εμείς. Και γι' αυτό, όπως και εκείνοι έτσι και εμείς, έχουμε κάθε συμφέρον και ενδιαφέρον να συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια. Και τα με Έθνη και εμείς, το Κοινοβούλιο, έχουμε μνημόνια συνεννόησης. Ήρθε η ώρα νομίζω να δημιουργηθεί ένα νέο σήμα ποιότητας, ένα νέο brand, label, το Διεθνές Masters στην Διερμηνία Συνεδρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει και διεθνείς γλώσσες, γλώσσες που δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να συμμετέχουν στο σήμα των Ευρωπαϊκών Masters. Και αυτό χωρίς να σημαίνει ότι θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας ή θα αφήσουμε κατά μέρο το European Masters. Είναι ο πρωτογενής μας. Όταν γίνεται ένα δεύτερο παιδί δεν αγαπάμε λιγότερο το πρώτο. Αντιθέτως. Περιμένουμε και το πρώτο παιδί να συμμετάσχει και να βοηθήσει το δεύτερο να μεγαλώσει καλά. Αυτή τη μεγάλη λοιπόν οικογένεια θέλουμε να την ανοίξουμε, αυτό και μόνο, προς, τα, προς όλα τα πανεπιστήμια είτε πρόκειται για γλώσσες ευρωπαϊκές είτε για γλώσσες μη ευρωπαϊκές, θέλουμε να ανοίξει ώστε να μπούμε όλοι σε μία οικογένεια με μόνο κριτήριο την ποιότητα. Όλοι δε εκείνοι οι οποίοι συμμερίζονται τις αξίες που καταγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης θα είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν σε αυτό το νέο σήμα. χωρίς να χαθεί το παλαιό σήμα, το παλαιό brand για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο, θα είναι και το ένα και το άλλο. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα μπορούν να συνεργάζονται στενά, χέρι-χέρι, με τα ρώσικα, κινέζικα, αραβικά πανεπιστήμια. Και ούτω καθεξής. Έχουμε αρχίσει να το μελετάμε. Θα χρειαστεί όμως πολύ περισσότερη μελέτη σε συνεργασία με εσά. Και σήμερα εγώ ρίχνω την ιδέα, τον όρο, την αρχή πάνω στην οποία θα στηθεί αυτό, αλλά σας καλώ να πάρετε, να κλείσετε ραντεβού και έχω ζητήσει από την Εμπρούντιρη Κέρι, η οποία ήδη είναι μέλος του δικτύου EMCI, αλλά και ως γλώσσα υποψήφιας χώρας, που δεν είναι ακόμα επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να αναλάβει τον συντονισμό για να θεσπιστεί αυτό το νέο δίκτυο, όπου θα συνδυαστούν οι ιδέες όλων των πανεπιστημίων, αλλά και όλων των, όπως λέμε σε καλά ελληνικά, των stakeholders, όλων των εμπλεκομένων φορέων. Υπάρχει μεγάλη γνώση και εμπειρία για γλώσσες που εμείς δεν έχουμε. Η Πάτη έχει εμπειρία όλων των γλωσσών του κόσμου, όλων των γλωσσών του κόσμου. Αν θυμάμαι καλά μου είχε πει ότι δεν θυμάται να υπήρξε μία γλώσσα του κόσμου που να μην χρειάστηκε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει στα διδρομία της. Και για όλους τους επικεφαλείς και τις υπηρεσίες διερμηνίας που θέλουν ένα και μόνο πράγμα, το επάγγελμα αυτό να προοδεύσει. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ποιότητα. Διότι αν δεν υπάρχει ποιότητα, τότε ναι, όντω είμαστε υπερβολικά ακριβοί. Κοστίζουμε πολύ, γιατί δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα. Εάν υπάρχει ποιότητα, το επάγγελμα έχει μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να αφήσω παρακαταθήκη αυτό το μήνυμα ελπίδας με τη δημιουργία αυτού του νέου δικτύου και ζητώ από την Εμπρού να θεσπίσει αυτό το δίκτυο με όλα τα πανεπιστήμια που ασφαλώς θα πρέπει να ζητήσουν ε, και από τους μη παρόντες ε, πριτάνης ή τις άλλες αρχές τους γνώμες και προτάσεις και βέβαια από τους επικεφαλείς των υπηρεσιών διερμηνίας όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό στο οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσουν να συμβάλλουν με την εμπειρία τους ο κάθε ένας και η καθημεία, ώστε κάθε γλώσσα να έχει τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Η διερμηνία είναι ένα οικουμενικό επάγγελμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα επάγγελμα με τεράστια κινητικότητα. Ένας διερμηνέας ο οποίος σήμερα είναι εγκαταστημένος με επαγγελματικά εκεί έδρα στην Ευρώπη μπορεί αύριο να εγκατασταθεί κάπου αλλού. Και μόνο εάν μοιραστούμε τα ίδια κριτήρια ποιότητας και τα ίδια κριτήρια επαγγελματικής διοντολογίας, όπως μας τα περιέγραψε η Πάτση νωρίτερα, Μόνο τότε θα έχει ένα μέλλον το επάγγελμά μας. Μόνο τότε θα είναι πραγματικά οικουμενικό. Σας ευχαριστώ θερμά που μου επιτρέψατε με την παρουσία σας. Να προωθήσω το όνειρο αυτό, το όραμα αυτό. Ελπίζω να το δούμε να ευμερεί με τον ίδιο τρόπο με το μωρό του Νοέλ και το δικό μου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς πολύ θερμά τους διερμηνείς, με τους οποίους, για τους οποίους, χάρη στους οποίους κατέστη δυνατόν όλο αυτό. Σας καλώ να χειροκροτήσετε τους εδώ παρόντες σήμερα, αλλά και εκείνους τους Γερμανείς που δεν είναι εδώ. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω να χειροκροτήσουμε όλοι θερμά όλους όσοι μας στήριξαν από το προσωπικό μας για την πιστοποίηση και την, ε, τις κάρτες εισόδου, που σας φρόντισαν οποτεδήποτε είχατε κάποιο πρόβλημα, κάποια ανησυχία, τους τεχνικούς μας που μας βοήθησαν με την ε, ε, με τα μηχανήματα, τον εκπρόσωπο της ε, υπηρεσίας των τεχνικών, ε, της τεχνικής υποστήριξης που, μας ήρθε, που ήρθε να μας βοηθήσει να ψηφίσουμε και εν τέλει και πάνω από όλους την Ιζαβέλα και τη Σουζάνε οι οποίες ήταν και οι άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε αυτό το έργο που εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο εργάζονται ακαταπώνητα. Δεν ξέρω αν ε, με καταριόντουσαν από μέσα τους με την ιδέα μου αυτή. Αλλά ε, εργάστηκαν ακαταπώνητα και θα ήθελα να σας πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ήμασταν σε διαρκή επαφή για το πόσες θέσεις θα έχουμε στην αίθουσα, για το ποιες θέσει θα έχουμε στο τραπέζι, ποιος θα κάτσει πού, Ποιο τελευταία στιγμή μα ενημέρωσε ότι θα έρθει, ποιο τελευταία στιγμή μα ενημέρωσε ότι θα έρθει. Και οι οποίε, σαν νεράιδε, διακριτικά και ήρεμα και ήσυχα φρόντισαν να γίνουν όλα σωστά. Για όλους αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους σας καλώ να χειροκροτήσετε θερμά. Enfin, je vais Εν τέλει, θα καλέσω εκείνη που παίρνει την ε, σκητάλη και θα με διαδεχθεί να έρθει εδώ και να δώσουμε και την ευκαιρία σε όποιον δεν είχε την ευκαιρία να τη γνωρίσει και να της μιλήσει, να γνωριστεί μαζί της. Αγνιέσκα Βάλτερ που ήταν ε, μέχρι τώρα στην πλευρά των Χριστών της Γερμανίας, τώρα θα αναλάβει το πιδάλιο για να σας μεταφέρω μια εικόνα που μου είχε μια μέρα μεταφέρει ένας επικεφαλής διερμηνέας και με χαροποίησε πολύ. Μου λέει πριν από χρόνια και λίγο λίγο μετά το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρδια. Ο, ο πλοίαρχος Κετίνο λοιπόν μου λέει αυτός ο διερμηνέας, ο κεφλής διερμηνέας μου λέει δεν ξέρεις πόσο ήσυχα αισθάνομαι που ξέρω ότι στο πιδάλιο βρίσκεται ένας πλοίαρχος που ξέρει που μας πάει. Της αφήνω ένα πλοίο το οποίο προχωράει στα νερά του, στρωμένα νερά, δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν θέλω να επενέσω αυτόν, αλλά είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί, που λειτουργεί πολύ καλά και είμαι πεπισμένη ότι όλοι σας θα τίνετε ευηγόνους και θα ξαναγυρίσετε σε ένα άλλο παγκόσμιο φόρουμ. Σας ευχαριστώ.